Καλημέρα σας. Είμαστε λίγο χαμένοι σε αυτή τη μεγάλη αίθουσα. Άρχεται η συνεδρίαση. Έχετε την ημερήσια διάταξη ε, μπροστά σας. Είναι όπως προβλεπόταν, αλλά έχει αλλάξει εδώ και δύο μέρες. Δεν θα ψηφίσουμε την έκθεση της κυρίας Φερχάιεν δεν θα την ψηφίσουν. Α, δεν υπάρχει διερμηνία προς τα αγγλικά. Πώς είναι δυνατόν. Φαίνεται ότι δεν λειτουργεί το σύστημα για κάποιο λόγο. Θα συνεχίσω στα αγγλικά λοιπόν. Η, η ημερήσια διάταξη βρισκόταν στην ιστοσελίδα μας εδώ και δύο ημέρες. Θα πρέπει όμως να μην γίνει η ψηφοφορία για τις δύο εκθέσεις Φερχάιεν, γιατί η Επιτροπή, η υπεύθυνη Επιτροπή δεν έχει ψηφίσει, γι' αυτό θέλουμε να την παρακολουθήσουμε εκ του Γιατί υπάρχουν πολύ σημαντικά και δύσκολα θέματα και νομίζω ότι θα πρέπει να κατανοήσουμε περί τίνος πρόκειται πριν αποφασίσουμε. Νομίζω ότι καταλάβατε, παρά τα κάκη στα αγγλικά μου. Άρα εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη, σημείο 3, έγκριση των πρακτικών. Δεν ξέρω κατά πόσο έχετε να πείτε κάτι πριν από τη λήξη της συνεδρίασης, διαφορετικά τα πρακτικά θα εγκριθούν. Υπάρχει τώρα αγγλική διερμηνία για να μην μιλάω αγγλικά όλη την ημέρα. Λοιπόν, η, τη συνεδρίασή μας ε, μπορεί να την παρακολουθήσει οποιοδήποτε από το διαδίκτυο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Έχουμε διερμηνία στο ίμιση των γλωσσών Όλες αυτές τις γλώσσες δεν τις έχουμε. Άρα οι Σλοβαίνοι για μία φορά είναι ευτυχείς διότι κατανοούν ακόμα και τα αγγλικά μου. Α, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Λέει η πρόεδρος στα γερμανικά πλέον. Λοιπόν, έχουμε ε, αγγλική διερμηνία. Ωραία. Συνεχίζω στα γερμανικά. Και περνάμε στον αθλητισμό. Ήταν πραγματικά το πιο σημαντικό θέμα από όλα. Κάθε ένα στην Ευρωβουλή πίστευε ότι έπρεπε να πει κάτι ή τα πάντα για τον αθλητισμό. Κατανοητό. Αλλά ήταν δύσκολο για τον συνάδελφο Φίσα όλα αυτά να τα εντάξει σε ένα κοινό πλαίσιο. Έχουμε λοιπόν την έκθεση του κυρίου Φίσας και ξέρετε ότι, πώς να το πω, κάποιες εκθέσεις είχαμε πιο πριν είχαμε και την έκθεση του Προέδρου της Ουγγαρίας, σημερινού Προέδρου της Ουγγαρίας για τον ρόλο του, του αθλητισμού στην εκπαίδευση και το μέλλον του επαγγελματικού ποδοσφαίρου και τώρα έχουμε το μέλλον, το, ε, οι άνθρωποι και ο αθλητισμός και στο μέλλον. Είναι το ότι βρίσκουμε τον αθλητισμό πάλι εδώ και ελπίζουμε ότι κάποιες πρόσθετες αρμοδιότητες για τον αθλητισμό θα δοθούν σε μας ο κύριος Φίσας στις 14 Ιουλίου παρουσίασε την έκθεσή του. 339 τροπολογίες είχαμε και έξι άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές ενεπλάκησαν και γνωμοδότησαν. Ωραίο αυτό, καλό. Λοιπόν, μπορώ να πω στον κύριο Φίσα ότι τον ευχαριστούμε βέβαια ότι έκανε τον κόπο να βρει ένα συνεκτικό πλαίσιο ως προς το εγγραφό του και ελπίζουμε στην ψηφοφορία σήμερα κάπως, πώς να το πω, θα είμαστε συνεκτικοί και εμείς να μην έχουμε πολλά πράγματα που θα αντιφάσκουν στην έκθεση και να μην έχουμε δυσκολίες στο τέλος να περάσουν τα μηνύματά μας προς τους πολίτες. Αν θέλει να πει κάτι ο Σαντιάγο, του δίνω τον λόγο. Παρακαλώ Σαντιάγο, έχεις τον λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Ντόρις Πακ. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέφους και ιδιαίτερα τους σκιώδεις εισηγητές για το θετικό πνεύμα συνεργασίας τους. Το πνεύμα να πετύχουμε ένα έγγραφο, όπως πολύ καλά είπες, να είναι συνεκτικό και υπέρ του αθλητισμού. Πρώτα απ' όλα είναι αυτονόητο <clears throat> σε σχέση με το σκιώδη εισηγητή της Σοσιαλιστικής και Δημοκρατικής Ομάδας, ε, Καταλήν, που συνεργάστηκε πολύ καλά μαζί μου και στον εισηγητή της Άλτε, Λίαμ Άλουορτ, που πάλι ήταν πολύ επικοδομητικό το πνεύμα συνεργασίας μας. Από πλευράς ε, Κλάρκιν, την υποστήριξη θέλουμε να τονίσουμε σε κάποια σημεία. Ήταν πολύ χρήσιμο όμως το ότι είχε κάποιες ιδέες που υπέβαλε για να βελτιωθεί το κείμενο. Επίσης να αναφέρω τον σκιώδη εισηγητή της ομάδας των Πρασίνων που δυστυχώς δεν παρίσταται. Κάνει την προεκλογική εκστρατεία στην Καταλωνία από πλευρά του. Και επίσης ε, την σκιώδη συγγήτρια της Γκουε, τη Μαρή Κριστίν Βερζά, που όπως ε, είπα συζήτησα και με αυτήν και όλους τους ευχαριστώ για το επικοδομητικό τους πνεύμα και είναι αυτονόητο επίσης και τη γραμματεία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπή, ιδιαίτερα τη Ρίτα που δούλεψε σκληρά και όλου του βοηθού θέλω να ευχαριστήσω και τους διαφορετικούς ε, συντάκτες γνωμοδότησης, διότι υπήρξαν βέβαια πολλές τροπολογίες. Θα έλεγα ότι οι απόψεις δεν ήταν τόσο ξεχωριστές και διαφορετικές. Ήταν όμως, θα έλεγα, πολλές και διαφορετικές και έπρεπε να γίνει η προσπάθεια να είμαστε συνεκτικοί, να έχουμε ένα κείμενο το δυνατόν πιο συνεκτικό. Εργάστηκαν και οι βοηθοί των διαφορετικών ευρωβουλευτών προς αυτό το σκοπό. Τους ευχαριστώ όλους λοιπόν και ελπίζω ότι θα έχουμε καλή ψηφοφορία και θα έχουμε στο τέλος ένα κείμενο που θα είναι θετικό για τον αθλητισμό. Αυτό αναμένεται από εμάς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Σαντιάγο. Ενώ μιλούσε ο φίλος σου Ιβαν, την φίλη του, Νεφενταλόβα την συνεχάρη για τα γενέθλιά της. Χρόνια πολλά και εμείς προσθέτουμε τη φωνή μας στα χρόνια πολλά κυρία συνάδελφε. Τόσο νέος έπρεπε να είναι κανείς άλλη μια φορά έτσι. Λοιπόν περνάμε στον πίνακα ψηφοφορίας τώρα. Τροπολογία 71 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Μια στιγμή. 79, 81 τώρα. 81 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε η 81. Συμβιβασμός 21 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Γυναικών 1 υπέρ, κατά, Αποχές απορρίφθηκε. Μια στιγμή, μια στιγμή. 20 λέει εδώ. Deutsche Amendment 126. Mein Gott, das ist ja furchtbar hier. Das ist big 162 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 2 γυναικών υπέρ γυναικών 19. Συγγνώμη πάλι. Πρέπει να προσέξω. Τώρα θα προσέχω από εδώ και πέρα. 19 γυναικών υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 84 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 91 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την 91 ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. 15 υπέρ, 12 εναντίον. Εγκρίθηκε. 158, 158 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Παρακαλώ να σηκώνετε τα χέρια σας γιατί αλλιώς δυσκολευόμαστε να δούμε τι γίνεται. Προφορική τροποποίηση 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Ποια είναι τώρα η 239 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 5 υπέρ. Όχι. 83 λέγεται. Πού φτάσαμε. Περίεργο αυτό που έχω εδώ. 83 τώρα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 86 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 88. Πώς είπατε εσείς. Δεν έχετε διερμηνία. Λοιπόν, προχωράμε. Είμαστε στην 88 τώρα, εντάξει. Σελίδα 5, έτσι, για να το βρείτε. 88 τροπολογία, σελίδα 5, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, 88 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 89 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε 90 υπέρ κατά θα ελέγξουμε ψηφίζουμε την 90 άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας αποτέλεσμα ισοψηφία 14-14 απορρίφθηκε συμβιβασμός 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 102 έτσι 102 τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 107 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Συμβιβασμός 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 123 από την άλλη σελίδα τώρα, στην άλλη σελίδα 123. 123 υπέρ, κατά, απόχες. Δεν το έχω εδώ. Α, τώρα το βρήκα. 123. Σε τρία τμήματα μάλιστα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, απόχες, εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, απόχες, θα ελέγξουμε. Δεύτερο τμήμα της 123 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας και αποτέλεσμα 15-15 ισοψηφία απορρίφθηκε. Τρίτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. 124 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. 126 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 23 υπέρ, Σας ζητώ συγγνώμη, τι κάνω σήμερα. 128 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 23 τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Πάμε στην 136 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 138 υπέρ κατά θα ελέγξουμε. 138 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 22 υπέρ, 8 εναντίον. Εγκρίθηκε. 139 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. 140 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. 141 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 8 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε προφορική τροποποίηση 2 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 135 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 151 υπέρ κατά και πάλι 151 υπέρ κατά δεν γίνεται, κυρία Μαρία Μπαντιά Κουτσέτ. Εσείς τι είσαστε υπέρ, κυρία Μα... Ε, Μπαντιά Κουτσέτ. 151 είπαμε. 151, τι γίνεται. 151 υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 155 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 156 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 159 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συμβιβασμός 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συμβιβασμός 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 172 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 173 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 175-176 ταυτόσημες υπέρ αυτών κατά, αποχές απορρίφθηκαν. Συμβιβασμός 12 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Πάμε στην τροπολογία 20. Πού είναι αυτή, εδώ, 20 μάλιστα. Ίνκο και Γιούρι υπέρ, κατά, αποχές απορρίφθηκε. 184 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. 185 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. 187 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 188 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε συμβιβασμός 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε πάμε στην τοπολογία ΙΜΚΟ 7 τοπολογία 7 από την άλλη σελίδα αυτή και Γιούρι υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 196 σε τρία τμήματα πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε δεύτερο υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε τρίτο υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 197 τροπολογία 197 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 198 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 200 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 201 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε συμβιβασμός 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 209 μια στιγμή από την άλλη σελίδα. 209. Ήβο. Εντάξει, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 211. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 212. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 213 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 215 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. Συμβιβασμός 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 221 Απ' την άλλη σελίδα και αυτή υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 222 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε προφορική τροποποίηση 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 224 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 225 Α, έχει αποσύρθει, εντάξει. Και η δική μου 226, 227 τώρα, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 229, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 230, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 231, υπέρ. Κατά, αποχές απορρίφθηκε. 232 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 233 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 237 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 238 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 240 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 200 συμβιβασμός 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 200 μια στιγμή συμβιβασμός 16 τώρα υπέρ κατά μια και πάλι υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 250 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε Προφορική τροποποίηση 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Πάμε στη 16 τώρα. Τι κάνουμε. Στην άλλη σελίδα. Δεν την βρίσκω. Εκεί κάτω, έτσι, Γιούρι 6, 6, 6, 6 υπέρ, συγγνώμη, κατά αποχές απορρίφθηκε. 234 υπέρ, κατά Συγγνώμη, λάθος. 254. 254. Πού είναι αυτό? Έχουμε τη Γιούρι 6 και την άλλη 6. Συγγνώμη. Συγγνώμη λοιπόν. 252 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 253 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε. 253 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα εγκρίθηκε. 22 υπέρ, 8 εναντίον. Περνάμε στην 254 υπέρ. Κατά αποχέσα απορρίφθηκε. Συμβιβασμός 17 υπέρ. Κατά αποχέσα εγκρίθηκε. Πάμε στην 18 μια στιγμή. Πού είναι η 18? Δεν την βρίσκω. Πού είναι. Μάλιστα, συμβιβασμός 18 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 265 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 266 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 267 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 269 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 270 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 272 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 273 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 274 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 275 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 277 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Πάμε στην 283 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 284 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Προφορική τροποποίηση 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Λίμπε 4 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την ΛΥΜΠΕ 4 ηλεκτρονικά. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 14-14. Η ισοψηφία απορρίφθηκε. 286 κατέπεσε. Τι είπατε εσείς. Χωρίς μικρόφωνο. Δεν ακούγεται. Δεν ακούγεται. Λοιπόν, Λίμπε, είπατε να επαναλάβουμε, εντάξει επαναλαμβάνουμε, Λίμπε 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Ξαναψηφίζουμε την 4. Υπέρ. Πέρας ψηφοφορίας. Τι είπατε? Πέρας ψηφοφορία. Four. Την 4 είπαμε. Και τώρα είναι πιο πολύ. 13-15. 13 υπέρ 15 εναντίον απορρίφθηκε. Περνάμε στην 288 υπέρ κατά αποχές. Απορρίφθηκε. Προφορική τροποποίηση 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 294 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 295 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 296 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 297 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 298 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 300 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 301 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 304 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 305 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 306 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 307 τώρα έτσι 307 λοιπόν υπέρ όχι Σαντιάγο, καταπίπτει λες. Αν το λες εσύ εντάξει. Δεν καταπίπτει. Αν λέει καταπέσει το ένα τμήμα δεν εγκρίθηκε το άλλο ναι. Πάμε στην 307 λοιπόν. Επειδή το ένα τμήμα δεν είχε εγκριθεί πιο πριν. Λοιπόν εντάξει. 307 λοιπόν υπέρ. Κατά. Εντάξει. Λοιπόν εγκρίθηκε. 308-309. Όχι. 310 λοιπόν. 310 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 311 και 312 ταυτόσημες υπέρ αυτών. Κατά αποχές απορρίφθηκαν. 313 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 315 και 316 υπέρ αυτών. Κατά αποχές απορρίφθηκαν 317 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 321 σε δύο τμήματα πρώτο υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε αν το πρώτο τμήμα λέει υιοθετηθεί και τα λοιπά 322 καταπίπτει 322 όμως τώρα υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Προφορική τροποποίηση 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 325 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 326 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 327 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 328 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 329, 330, 31 ταυτόσημες υπέρ αυτών κατά αποχές απορρίφθηκαν. Συμβιβασμός 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Η 338 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 339 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Η 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Η 30 υπέρ. Α, τι λέω. Πού πήγα στην 30. 10, 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 13 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 15 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 22, 23, 24, 25 υπέρ αυτών κατά αποχές εγκρίθηκαν 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Προφορική τροποποίηση 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 28 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 29 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 31 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 32 υπέρ κατά αποχές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 κατά αποχές εγκρίθηκε 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε προφορική τροποποίηση 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 51 υπέρ κατά και πάλι υπέρ 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 53 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 54 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε περνάμε τώρα στην 60 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συμβιβασμός 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 65 υπέρ υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 67 σε τρία τμήματα πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε δεύτερο υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε τρίτο υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 69 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Προφορική τροποποίηση 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 6 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. μπορούμε να πάμε από το, να τις ψηφίσουμε και τις 12 από, από κοινού 1 έως 12 συμφωνείτε από κοινού ωραία ποιος είναι υπέρ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 κατά αποχές απορρίφθηκαν Οι 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε Οι 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 19 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε Οι 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε Τρία υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε Ένα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε Ένβη, η γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Ένβη. 4, 5, 6, 7 από κοινού γίνεται. 4, 5, 6, 7 ομού. Όχι 4 λοιπόν. Υπέρ. 4 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 5 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 7 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 8 όχι λάθος 7 τώρα έχετε 7 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε Τι λέει εδώ, αν υιοθετηθεί η έξι ο συμβιβασμό, το δεύτερο τμήμα τι καταπίπτει. Δεν πρέπει να ψηφίσουμε λοιπόν. 14 τώρα. Τι είπατε. Παρόλα αυτά θα ψηφίσουμε, είπατε, εντάξει, 11 λοιπόν, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. Η 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Η 1 καλύπτεται λέει από την άλλη, οπότε εντάξει, δεν θα ψηφιστεί. Τρομερό. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο ευγενικέ προ εμά όλε οι άλλε κοινοβουλευτικέ επιτροπέ να ψηφίζουν έτσι όπω εμεί ψηφίζουμε και δεχόμαστε. Είμαστε όμω πολιτιστικά ιδιαίτερα αναβαθμισμένοι και το κάνουμε εμεί αυτό. Ήμκο τώρα, τροπολογία 1. Δεν θα ψηφιστεί λέει. Ατυχία 2. <laughs> Κατά αποχέ εγκρίθηκε. 3. Υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίθηκε. Τι κάνουμε τώρα. Πέντε πέντε λοιπόν υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 8 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 9 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 13 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 14 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 16 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε δεν θα ψηφιστεί το α το β, β υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Σ Γ υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. D δεν θα ψηφιστεί. Εντάξει, η γνωμοδότηση της Γιούρη, η 4 υπέρ, κατά αποχές απορρίφθηκε. Το α της Γιούρη υπέρ, κατά αποχές απορρίφθηκε. Το C Γ της Γιούρη υπέρ, κατά αποχές απορρίφθηκε. Η γνωμοδότηση τη Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, ΛΥΜΠΕ, μια στιγμή, προφορική τροποποίηση 11 πρώτα, υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίθηκε. 8 της ΛΥΜΠΕ, υπέρ, κατά, αποχέ, απορρίφθηκε. 9 υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίθηκε. 13 υπέρ, κατά, αποχέ, απορρίφθηκε. Τώρα η Επιτροπή Γυναικών, η γνωμοδότηση τη Επιτροπή Γυναικών. Για όνομα του Θεού, τι γίνεται εδώ. Μάλιστα, ωραία. Η 4 <clears throat> υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 6 υπέρ κατά θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την 6 άρχεται η ψηφοφορία. 6 της Επιτροπής Γυναικών η 6 πέρας ψηφοφορίας γιατί γελάτε όλοι έτσι χαζά 19 εναντίον 11 υπέρ απορρίφθηκε η 7 γυναικών υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 8 υπέρ κατά <laughs> αποχές απορρίφθηκε. 10 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την 10 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 15-15 ισοψηφία απορρίφθηκε. 11 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 13 υπέρ κατά θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την 13. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 19 αντίον 11 υπέρ απορρίφθηκε. 14 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 17 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 21 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την 21. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 19 αντίον 11 υπέρ απορρίφθηκε. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την 1. Άρχεται πέρας ψηφοφορίας αποτέλεσμα 16 υπέρ 14 εναντίον εγκρίθηκε Θεέ μου μεγάλη επιτυχία οι δύο υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε ψηφίζουμε την 2 άρχεται πέρας ψηφοφορίας αποτέλεσμα 13 εναντίον 17 υπέρ εγκρίθηκε η 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 5 υπέρ κατά αποχές έλεγχος <clears throat> άρχεται η ψηφοφορία ψηφίζουμε την 5 πέρας ψηφοφορίας 14 ε, εναντίον 16 υπέρ εγκρίθηκε δεν χρειαζόταν και να το κοιτάξουμε αλλιώς τελική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία τελική ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας 28 υπέρ, 2 εναντίον. Συγχαρητήρια. Θα σε ευχαριστώ Σαντιάγο. Ήταν δύσκολο έργο αυτό που είχες επομιστεί. Αποκινούμε τους γνωμοδότες ε, συντάκτη γνωμοδότη και σκιώδης συζητητές. Επίσης ε, και Μακλάκιν θέλω να ευχαριστήσω. Υπήρξε μεγάλη συμφωνία. Έτσι ή όχι. Είπα εσείς 80% εντάξει 80 όχι πιο πάνω εντάξει έστω καλό και αυτό. Περνάμε τώρα στην έκθεση Σάκε. Η κυρία Σάκε δυστυχώς δεν παρίσταται. Παρόλα αυτά θα ψηφίσουμε, έτσι. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Τάκουλα, έχεις κάτι να πεις από την κυρία Σάκα ή όχι. Γίνεται και χωρίς παρέμβαση. Εντάξει, ωραία. Ξεκινάμε, ψηφίζουμε. Πολύ ωραία. Για την ανταγωνιστική ενιαία ψηφιακή αγορά. Μάλιστα, σημαντικό θέμα Το Συμβασμός 1, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 1. Όχι, Απ' την άλλη σελίδα. Προφορική τροποποίηση 1 υπέρ κατά. Μάλιστα, θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Προφορική τροποποίηση 1. Σελίδα 2. Αυτή ψηφίζουμε. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Μαρή Κριστίνα Βερζιά. 16 εναντίον 12 υπέρ απορρίφθηκε. Μάλιστα. Περνάμε στην τροπολογία 7 σε δύο τμήματα. Πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Δεύτερο υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα της 7 άρχεται πέρας ψηφοφορίας και αποτέλεσμα 18 εναντίον 12 υπέρ απορρίφθηκε 9 τροπολογία υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε συμβιβασμός 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε τροπολογία 15 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την 15. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 22 υπέρ, 7 εναντίον εγκρίθηκε. 16 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 17 υπέρ, κατά, αποχές. Θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την 17. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 15-15 ισοψηφία απορρίφθηκε. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 20 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την 20 άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 15 υπέρ 14 εναντίον εγκρίθηκε. 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 23 υπέρ κατά, αποχές, θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την 23, άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 13 υπέρ 16 εναντίον απορρίφθηκε. 24 τώρα και 25 υπέρ αυτών κατά αποχές απορρίφθηκαν. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 22 καταπίπτει 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 29 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 30 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε ψηφίζουμε την 30 άρχεται πέρας Αποτέλεσμα 16 υπέρ 14 εναντίον εγκρίθηκε. 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τι είπατε? Χωρίς μικρόφωνο δεν ακούγεται. 33. Ναι, σε αυτή θα φτάσω τώρα. Δεν είχα φτάσει εκεί. 33 λοιπόν υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 35 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 34 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 36 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε ψηφίζουμε την 36 άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας 19-11 εγκρίθηκε 37 υπέρ κατά αποχές Μα τι γίνεται, θα ελέγξουμε πάλι. Άρχεται η ψηφοφορία, ψηφίζουμε την 37, πέρας ψηφοφορίας. 16-13 απορρίφθηκε, 39 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 38 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 40 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 41 υπέρ, κατά, αποχές απορρίφθηκε 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 43 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε ψηφίζουμε 43 άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας τώρα και αποτέλεσμα 14 εναντίον 16 υπέρ εγκρίθηκε 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 47 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε περνάμε στην τελική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά πέρας ψηφοφορίας και αποτέλεσμα η κυρία Σάρκε με καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή με 30 ψήφους κέρδισε, εγκρίθηκε η έκθεση. Συγχαρητήρια, <laughs> όποια και να είναι. Σίγουρα μπροστά σε έναν υπολογιστή, εντάξει, πολύ ωραία. Τελειώσαμε. από πλευράς του συναδέλφου Μπερλίνγκερ μόλις έφτασε. Πολύ ωραίο το ότι ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Περνάμε τώρα στο σημείο 11. Συνεισφορά των ε, ευρωπαϊκών θεσμών στο 8 ευρωπαϊκή θεσμική, ε, θεσμικά όργανα, ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα στην της προόδου της διαδικασίας της Μπολόνια. Ξέρουμε ότι στην αρχή ήταν διακυβερνητικό εγχείρημα. Εμείς ως Ευρωκοινοβούλιο δεν εμπλεκόμαστε. Εμείς όμως πάντα υφιστάμεθα τις επικρίσεις και γι' αυτό πριν από τρία χρόνια είχαμε και μια έκθεση που συντάχθηκε για την διαδικασία Μπολόνια. Θεωρήθηκε αναγκαίο τώρα εκ νέου να συνταθεί μια νέα έκθεση γιατί οι κυβερνήσεις συμφώνησαν να βελτιώσουν κάτι στην στη διαδικασία Μπολόνια. Ο κύριος Μπερλιγκουέρ τα είδε αυτά από κοντά και μια και είχαμε την σύνοδο το 2010 που θα είχαμε βελτιώσεις ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε παρακαλώ τον κύριο Μπερλιγκουέρ να παρουσιάσει την έκθεσή του στις 23 θα έχουμε το σχέδιο έκθεσης που θα μας υποβληθεί στις 21 Δεκεμβρίου στη συνέχεια θα ψηφίσουμε προς έγκριση ο συνάδελφος Μπερλιγκουέρ παρακαλώ να μας δώσει την εισαγωγή του και να παρουσιάσει τις απόψεις του Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία για να συνοψίσω την, ε, το σκοπό της πρωτοβουλίας και συνεπώς και του κειμένου της ε, πρότασης ε, γνωμοδότησης ε, για το ρόλο των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων στην εδραίωση και την πρόοδο της διαδικασίας της Μπολόνια. Γνωρίζουν οι συνάδελφοι ότι το μήνα Απρίλιο του χρόνου θα λάβει χώρα η συνεδρίαση η διακυβερνητική συνεδρίαση που λαμβάνει χώρα κάθε δύο χρόνια και που πλέον αποτελεί θεσμό σχέση με την ενημέρωση των στόχων της υλοποίησης της διαδικασίας της Μπολόνια. Θα λάβει χώρα στο Βουκουρέστι. Η πρωτοβουλία λοιπόν του Κοινοβουλίου έρχεται σε μια στιγμή όπου τα πράγματα κινούνται ε, προς, ε, σε αυτό το τομέα. Η απόδειξη αυτής της κινητικότητας ήταν μια συζήτηση που έγινε σε αυτήν εδώ την Επιτροπή πολύ, ε, σε βάθος ε, και, βάση της, ε, και έγινε βάση της πρωτοβουλίας του Προέδρου που ζήτησε την εκπόνηση μιας μελέτης Και θα ήθελα να αναφέρω επίσης ότι πρόσφατα έλαβε χώρα η ολοκληρωμένη συζήτηση για τη διατύπωση των στόχων της Ευρώπης 2020 όπου υπενθυμίζεται η θεματολογία και επίσης οι διαφόρες πρωτοβουλίες της Κομισιόν για τον εξυγχρονισμό των πανεπιστημίων, μελλοντικά προγράμματα ε, ε, εκπαίδευσης, παιδείας και πολιτισμού και η ενημέρωση που είχαμε πρόσφατα. Έτσι δίνεται λοιπόν ιδιαίτερη ε, προσοχή στην κινητικότητα ως ε, κεντρικό θέμα, ως δικαίωμα στην Ευρώπη μας και προς υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων. Ποιος είναι ο σκοπός της πρότασης έκθεσης ε, που σας παρουσιάζω. Σκοπός είναι να αξιολογήσουμε αυτή τη διαδικασία η αποδοχή της διαδικασία της Μπολόνια ως θεμελιώδου στοιχείο για τη μεταρρύθμιση των πανεπιστημίων στην Ευρώπη θα πρέπει να χαρακτηριστεί περισσότερο ως δυναμική διαδικασία. Στο εσωτερικό του λοιπόν θα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τι ακριβώς αξίζει από όσα έχουν υλοποιηθεί μέχρι αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να δούμε την εγκυρότητα του γενικότερου στόχου και Επίσης, ε, από την άλλη άποψη, ποια ήταν τα σημεία, ας τα εμπόδια, τα σημεία συμφόρησης, ε, όπως τα αναφέρω στο συνοδευτικό έγγραφο της έκθεσης, και δηλαδή τα ελλείψεις ε, που έχει οποιαδήποτε μεταρρύθμιση και ειδικότερα η δική μας θα πρέπει καταρχάς να αναδείξουμε τον βαθύτερο στόχο. Ο βαθύτερος στόχος είναι ότι οι νέοι, τα παιδιά της Ευρώπης που εγγράφονται σε ένα πανεπιστήμιο οποιοδήποτε κράτους μέλους έχουν σήμερα το δικαίωμα όχι μόνο και την ανάγκη που προκύπτει από την εσωτερική μας αγορά να αποκτήσουν ένα πανεπιστημιακό πτυχίο το οποίο θα ισχύσει ολόκληρη την επικράτεια της Ευρώπης. Δεν θα πρέπει πλέον να υπάρχουν αυτόνομοι τίτλοι σπουδών στην Ευρώπη. Φυσικά η επιστημονική, πολιτισμική βάση ξεκινάει, βασίζεται στην εθνική παράδοση των κρατών μελών, ωστόσο η εγκυρότητα θα πρέπει να ισχύει σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό μας θέτει προβλήματα, επειδή αυτή τη στιγμή όσοι συμμετέχουν στη διαδικασία της Μπολόνια είναι αυτή τη στιγμή είναι 47 κράτη-μέλη σε σχέση με τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι έχει τεράστια επιτυχία. Ε, και εκτός Ευρώπης ο πρωταρχικός στόχος παραμένει να έχουμε ένα πανεπιστήμιο κατά, γενικό, ε, γενική έννοια ευρωπαϊκό που θα αποτελείται από τα επιμέρους κράτη-μέλη και τις δικές τους παραδόσεις. Η εγκυρότητα του τίτλου που παρέχεται αποτελεί πλέον ε, ε, υποχρέωση για την οικοδόμηση της Ευρώπης σήμερα στην ε, δημοκρατία των γραμμάτων όπως ε, λεγόταν στο τομέα των διαφορετικών επιστημών στους οποίους αντιστοιχούν οι διάφοροι τίτλοι σπουδών η αγορά εργασίας απαιτεί όλο και περισσότερο να υπάρχει εσωτερική κινητικότητα και δυνατότητα εφαρμογής εργασίας στον τομέα του καθενός οπουδήποτε τα κράτη-μέλη σήμερα και τα πανεπιστήμια δεν έχουν δεσμευτεί επαρκώς ώστε αυτή η, η, υποχρέωση κατά κάποιο τρόπο να μας βοηθήσει να επιτύχουμε το αποτέλεσμα. Η διαδικασία είναι πολύ αργή, δεν υπάρχουν διασφαλίσεις ώστε να εφαρμοστεί αυτή η διαδικασία σε βάθος. Ποιος είναι, ποια είναι τα κοινωνικά αίτια, όχι μόνο πολιτισμικά και επαγγελματικά. Τα αίτια είναι ότι σήμερα, οικοδομώντας μια ευρωπαϊκή ηθαγένεια, εμείς χρειαζόμαστε και μια πανεπιστημιακή ευρωπαϊκή ηθαγένεια, μια πολιτισμική ηθαγένεια, επαγγελματική ηθαγένεια ευρωπαϊκή. Αυτό είναι ένας τους πρωταρχικούς στόχους που πρέπει να έχει η Ένωση και μαζί της ε, τα κράτη-μέλη ένας πρωταρχικός στόχος τον οποίο δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε. Αποτελεί κινητήριο μηχανισμό. Θα πρέπει να έχουμε την αίσθηση, την ε, επίγνωση ότι τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κρατών μελών θα πρέπει να έρουμε τα εμπόδια και τις δυσκολίες που αντικειμενικά αντιτίθενται σε μια, σε μια αλλαγή σαν αυτή που είναι από τις πιο ε, βαθιές αλλαγές που έχουν λάβει χώρα στην Ήπειρό μας. Σήμερα οικοδομούμε μια Ευρώπη, έναν ευρωπαϊκό χώρο ανώτατης ε, εκπαίδευσης, το EHEA. Ενώ ταυτόχρονα ε, οικοδομούμε τον ευρωπαϊκό χώρο έρευνας. Ε, συνεπώς, στους τομείς ε, εξειδικευμένης έρευνας υπάρχει απέτηση για ευρωπαϊκή παιδεία, όχι μόνο ως υποχρέωση. Βλέπω ότι η Ευρώπη έχει αποφασίσει, ακόμη παρότι λίγο δειλά και με πολύ αργά βήματα, έχει αποφασίσει να πρωταγωνιστήσει η ίδια η Ευρώπη δηλαδή να διαδραματίσει ένα ρόλο στην ανώτερη εκπαίδευση, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στην έρευνα. Φυσικά ο πρωταρχικό ρόλο θα διαδραματιστεί από τα κράτη-μέλη. Κανεί δεν αμφισβητεί κάτι τέτοιο. Ήδη οι συνθήκε το λένε καθαρά και εμεί δεν έχουμε καμία βούληση να παραβιάσουμε τι συνθήκε. Ωστόσο, όλα δείχνουν ότι ακόμη και αυτή τη στιγμή στην ευρωπαϊκή νομοθεσία υπάρχει ένα προφίλ ε, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας και αυτό το προφίλ αφορά περισσότερο το ρόλο παρά τις ε, ικανότητες. και αποτελεί κομμάτι της ζωής μας. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ένα από τα κεντρικά σημεία αυτού του αποτελέσματος είναι η αμοιβαία αναγνώριση της εγκυρότητας των τίτλων σπουδών μεταξύ των χωρών και μεταξύ πανεπιστημίων. Αυτό είναι ένα από τα ενδιάμεσα βήματα που θα οδηγήσουν στον τελικό στόχο, στην αυτόματη αναγνώριση στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια παρότι αυτό δεν θα έλεγα βέβαια όνειρο αλλά είναι ένας ε, στρατηγικός στόχος ε, όχι τόσο τακτικός η αμοιβαία αναγνώριση. Θα σας δώσω το παράδειγμα της ε, χώρας μου, η Ιταλία, η οποία ανησυχεί για την αναγνώριση των τίτλων μέσα στην ίδια την Ιταλία δεν μπορεί αυτή να προωθεί την αναγνώριση των τίτλων των άλλων χωρών. Θα πρέπει να υπάρξει κάτι υπερεθνικό, το οποίο θα ευνοήσει την κατάκτηση αυτού του αποτελέσματος. Το να λέμε λοιπόν ότι εδώ μιλάμε μόνο για αρμοδιότητα των κράτων μελών, σημαίνει ότι δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τον ευρωπαϊκό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Γι' αυτό το λόγο προσπαθούμε να λάβουμε αυτή την απόφαση. Με μεγάλη ελπίδα και με μεγάλη χαρά διάβασα ότι η Κομισιόν, σύμφωνα με τα λόγια της Επιτρόπου, της κυρίας Βασιλείου, στον εξυγχρονισμό των πανεπιστημίων αλλά και στην ανακοίνωσή της ΑΝΤΟΚ ασπάστηκε αυτή τη θέση. Αυτό σημαίνει ότι σήμερα τα θεσμικά όργανα της Ευρώπης αρχίζουν να συγκλίνουν προς μια κατεύθυνση όπου μας οδηγούν ε, τα γεγονότα. Πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Σίγουρα ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε είναι, βασίζεται σε μικτές ενδείξεις ε, ε, τόσο όσον αφορά την νομοθεσία αλλά και όσον αφορά και τα κίνητρα υποστήριξης της διαδικασίας της Μπολόνια. Σήμερα περισσότερο από χθε θα πρέπει να πλαισιωθεί στο ε, τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα πρέπει να γίνει αυτός ο χώρος ένα ενιαίο κομμάτι. Αυτό είναι το βασικό βήμα το οποίο θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε πιο αποφασιστικά. Όλα αυτά όπως φυσικά είπα θα πρέπει να αναδείξουν το ίδιο το όνομα της διαδικασίας. Διαδικασία σημαίνει από κάτω προς τα πάνω, όχι μόνο από πάνω προς τα κάτω δεν μπορούμε να το αναθέσουμε, δεν μπορούμε να αναθέσουμε μια τέτοια διαδικασία μόνο στις διετής ε, συνεδριάσεις των Υπουργών Παιδείας ε, επί του θέματος, ούτε μόνο στις ε, διασκέψεις κορυφής των κρατών και των κυβερνήσεων, ούτε μόνο στις συνεδριάσεις των Πριτάνεων από διάφορες χώρες που ήδη λαμβάνουν χώρα. Δεν μπορούμε να αναθέσουμε ένα τέτοιο έργο μόνο στις διασκέψεις κορυφής. Θα πρέπει να αποτελέσει καθημερινή διαδικασία ολόκληρου του ακαδημαϊκού σώματος και του φοιτητικού σώματος στην Ευρώπη. Εμείς δεν έχουμε καταφέρει να επιτύχουμε τη συμμετοχή αυτών των σωμάτων. Δεν έχουμε καταφέρει να τους κάνουμε να αισθανθούν υπεύθυνοι. Δεν τους έχουμε ενθαρρύνει και να, δεν, έχουμε, τους έχουμε δώσει κίνητρα που πάντα ενθαρρύνουν ε, ε, κινήσεις αυτού του τύπου δεν έχουμε καταφέρει να αποδείξουμε ότι μια τόσο σημαντική μεταρρύθμιση θέτει σε συζήτηση την ίδια μεθοδολογία, την ίδια την τακτική. Διότι ας πούμε ότι διδάσκεται σε τρία χρόνια είναι διαφορετικό από ότι διδάσκεται σε πέντε χρόνια και αυτό αποτελεί επανάσταση τακτικής και αλλάζει τον τρόπο που οι διάφορες χώρες ε, βλέπουν τα πράγματα. Εγώ από της, προερχόμενος από χώρα του Νότου αισθάνομαι αυτή την καθυστέρηση σε σχέση με τις χώρες του Βόρα. Και αυτή τη διαφορά που υπάρχει στην Ένωσή μας θα πρέπει λοιπόν να υπογραμμίσουμε αυτή την εκπαιδευτική και διδακτική μεθοδολογία δεν έχουμε καταλάβει ότι χρειάζεται μια πιο βαθιά κοινωνική ευαισθησία η οποία να στην οποία να συμμετέχουν ε, ο κόσμος των πανεπιστημίων και των φοιτητών που για κάποιους λόγους ακόμα βρίσκεται στο περιθώριο. Η Ευρώπη θα πρέπει να μπορεί να αξιοποιήσει όλο, όλη την ευφυΐα όλων των νέων που υπάρχουν ε, και όχι μόνο ε, των προνομιούχων. Αυτές είναι οι δύο πτυχές, μία καθαρά πολιτισμική και εκπαιδευτική, η άλλη κοινωνική και αυτές οι πτυχές καθιστούν τον ευρωπαϊκό χώρο της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ε, έναν στόχο φιλόδοξο που θα πρέπει να υποστηρίξουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Θα σας ε, δώσω μια εικόνα των πρακτικών σημείων που ε, επισημένονται και που έχουν λάβει προσοχή στο παρελθόν αλλά όχι επαρκώς. Όπως είπα ο πρώτος στόχος είναι η αναγνώριση των τίτλων σπουδών οπουδήποτε. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπογραμμίσουμε την αξία του βασικού δικαίου κινητικότητας. Του βασικού δικαιώματο συγγνώμη, κινητικότητα. Και αυτό δεν μπορεί να επιβληθεί μόνο με νόμους. Ας δούμε το παράδειγμα του Εράσμους, ένα από τα πιο επιτυχή έργα στην Ευρώπη ε, επηρέασε εκατοντάδες χιλιάδες από τα παιδιά μας. Παρότι σήμερα βρισκόμαστε σε ένα σημείο κρίσης, ε, επειδή είχε σχεδιαστεί με σκοπό να στέλνουμε έναν φοιτητή από το σπίτι του σε ένα άλλο κράτος μέλος, ε, σήμερα υπάρχει η φιλοδοξία να υπάρχει το Erasmus 3.2. Η χώρα υποδοχή σήμερα θα πρέπει να παίξει κάποιο ρόλο και αυτήν θα πρέπει να υποστηρίξουμε. Η διδακτική υπηρεσία θα πρέπει να λειτουργήσει περισσότερο από το δικαίωμα μετακίνησης. Αυτό μας δείχνει ότι υπάρχει μια ε, πολιτική αλλαγή που θα πρέπει να επιβάλλουμε. Όχι δηλαδή να δίνουμε σημασία στην κίνηση προς την άλλη χώρα, αλλά ε, στη χώρα που ε, υποδέχεται τους φοιτητές από μια άλλη χώρα. Εδώ παίζει ρόλο η αναγνώριση των ε, τίτλων σπουδών. Ε, καταλαβαίνω ότι μια χώρα μπορεί να μην δεχθεί να εργαστεί ως γιατρός εκεί ένα άτομο που έχει λάβει τίτλο σε άλλο κράτος μέλος και φυσικά ίσως να μην μπορεί να εμπιστευτεί έναν επαγγελματία που έχει λάβει ε, πτυχίο αλλού. Ίσως λοιπόν να υπάρχει κάποιο πρόβλημα εμπιστοσύνης όσον αφορά την ποιότητα. Γι' αυτό λοιπόν, για να μπορέσει να υπάρξει αμοιβή εμπιστοσύνη, θα πρέπει να υπάρχει έλεγχο, επαλήθευση. Η επαλήθευση αυτή θα πρέπει να είναι κάτι καθημερινό, όχι κάτι ε, περιστασιακό το οποίο θα λαμβάνει χώρα όσον αφορά τα αποτελέσματα της παιδείας. Εμείς ε, στην Ευρώπη αυτό δεν το έχουμε κίνητρα λοιπόν ε, ε, η νομοθεσία, οι θεσμικές αρχές θα πρέπει να προβλέψουν σε κάθε κρατος μέλος ακόμη και στο επίπεδο του ε, Μητρώου Αξιολόγησης Ικανοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο η πολιτική επαλήθευσης και αξιολόγησης είναι απολύτως απαραίτητα. Το επόμενο στοιχείο είναι η απασχολησιμότητα. Τι δουλειά κάνουν οι πτυχιούχοι έχει, υπάρξει, έχει συζητηθεί το τριετές πτυχίο. Τομείς όπου δεν έχει γίνει κατανοητό περί τίνος πρόκειται και σε άλλους τομείς λειτουργεί. Σήμερα μας λένε διάφορες έρευνες ότι οι πιο προηγμένοι οικονομικοί τομείς έχουν κατά κάποιο τρόπο καταγράψει την ανάγκη τριετούς πτυχίου επειδή ο πλούτος και η διάρθρωση της αγοράς εργασίας ε, δεν αφορά πλέον εκπαίδευση σε ένα μόνο ε, επάγγελμα, αλλά σε πολλά επαγγελματικά επίπεδα, τα οποία περιλαμβάνουν περισσότερα επίπεδα ε, εκπαίδευσης. Ε, έχουμε ήδη στατιστικά στοιχεία τα οποία μας λένε ότι οι χώρες που έχουν συνεργαστεί σε ένα συνδυασμό ζήτησης και προσφοράς μεταξύ και σε μια συνεργασία μεταξύ του κόσμου της αγοράς και του κόσμου της παιδείας έχουν καταφέρει να προσαρμόσουν αποτελεσματικά ακόμη και τα τρίτη πτυχία. Άλλες χώρες αντιθέτως έχουν αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα με απλή... Ε, ε, κατά περίπτωση χρειαζόμαστε λοιπόν μια στάση επικοδομητική και όχι να αξιολογούμε τα καλά και τα κακά θα πρέπει να το κάνουμε όλο αυτό επικοδομητικά επειδή ε, χτίζεται η Ευρώπη μέρα με τη μέρα. Και το ζήτημα της αποσχολησιμότητας έχει γίνει αποφασιστικό από αυτή την άποψη. Η άλλη πτυχή είναι η ευελιξία των προγραμματών σπουδών. Συχνά σε πολλές ε, χώρες έχουμε πολύ αυστηρά προγράμματα σπουδών και γι' αυτό είναι τόσο δύσκολο να τα συγκρίνουμε. Κανείς δεν έχει σκεφτεί να υπάρχει ένα ενιαίο πρόγραμμα σπουδών στην Ευρώπη. Αυτό είναι δύσκολο πολιτισμικά και επιστημονικά. Αυτό είναι ένα επιστημονικό λάθος. Αλλά στο να υπάρχει ένας εσωτερικός πυρήνας στο πρόγραμμα το οποίο να έχει μία ε, κοινή ισχύ ε, να αφορά κάποια βασικά στοιχεία και εκεί να προστίθενται όλα τα διάφορα στοιχεία που οφείλονται στους διάφορους πολιτισμούς και στις διάφορες παραδόσεις αυτό μπορεί να γίνει. Υπάρχει ήδη με άλλες πρωτοβουλίες, υπάρχουν ήδη λύσεις οι οποίες έχουν δοκιμαστεί πειραματικά. Εκεί θα πρέπει να ενθαρρύνουμε και να δώσουμε κίνητρα. πριν φτάσουμε σε κάποιο κοινό τίτλο ή σε μια κοινή πούμε, αναγνώριση για κάθε τομέα, η ιδέα του να πολλαπλασιάσουμε τα joint degrees, δηλαδή τις διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες, ε, από διάφορους επιστημονικούς τομείς ή από διάφορα πανεπιστήμια θα μπορούσε να αποτελέσει μία εδώ που θα μας οδηγήσει σε κάποιο αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι χονδρικά πιστεύω ότι σήμερα με θετικό και επικοδομητικό τρόπο ε, μπορούμε να προχωρήσουμε στο μέλλον Learning Centered System. Αυτή η εφαρμογή μπορεί να μας χρησιμεύσει. Ξεκινάμε δηλαδή με βάση τη ζήτηση και όχι την προσφορά. Δίνοντας την τρίτη αποστολή μια έννοια του πανεπιστημίου που θα προσαρμόζεται σε μια κοινωνία βασισμένη στην γνώση αλλά και στις ε, τεχνολογίες ε, πληροφορίας ε, και στην ευρύτερη εφαρμογή της εκπαίδευσης επίσης. Πρώτα απ' όλα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στη Μεσογεία και στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης επειδή εκεί υπάρχουν ήδη μορφές της διαδικασίας της Μπολόνια όπου έχουν συμπεριληφθεί αυτά τα κράτη-μέλη και τα πανεπιστημιακά συστήματα. Σκέφτομαι τη Βόρειο Αφρική που, ε, όπου, που συμμετέχει και σκέφτομαι επίσης και τις ανατολικές χώρες. Μέσω αυτών των προσεγγίσεων προσπαθούμε μέσω της έκθεσης να φτάσουμε σε κάποιο σημείο υλοποίηση και παγίωσης ε, του ευρωπαϊκού χώρου ε, βάθμιας εκπαίδευσης. Ευχαριστώ. Ένας καθηγητής ομίλησε, όμως που δεν ζει σε ένα λαβάστρινο πύργο, αλλά που ξέρει από την καθημερινή ζωή ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα. Ξέρω και στην Ιταλία σε πανεπιστήμια το έχω βιώσει, αυτό το έχω ζήσει. Έχει υψηλό σεβασμό που απολάβει και η Ιταλία και αυτός και χαίρομαι που το έκανε τόσο διεξοδικά. Τα προβλήματα ποτέ ουσιαστικά δεν αντιμετωπίστηκαν στο παρελθόν. Και αν σήμερα, δέκα χρόνια μετά την έναρξη, μια τέτοια περιγραφή, μια περιγραφή πρέπει να δοθεί. Αυτό δείχνει πόσο ερασιτεχνικό ήταν το επίπεδο της διακυβερνητικής διεργασίας, διακυβερνητικής προσέγγισης. Και αυτό επειδή οι κυβερνήσεις ζουν υπό τη δαμόκλειο σπάθη της επικουρικότητας και δεν γίνεται κάτι διαφορετικό. Θλιβερό είναι αυτό βέβαια. Ευχαριστούμε θερμά συνάδελφε Μπέρλιγκουερ. Δώσατε πολλά ερεθίσματα για μια συζήτηση που θα διεξαχθεί τώρα. Η κυρία Κάμε Εύερτ παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε για αυτά που μόλις είπατε. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά βέβαια. Ο κύριος Μπερλιγκουέρ πάρα πολλές πτυχές ανέφερε που νομίζω όλοι, όλες μας συγκινούν και μας κάνουν να θέλουμε να αντιδράσουμε. Οι στόχοι που περιγράφηκαν από τη διαδικασία της Μπολόνια εξακολουθούν να είναι σωστοί. Μόνο που διαπιστώνουμε ότι 10 χρόνια μετά την έναρξη αυτής της διαργασίας της Μπολόνια αυτοί οι στόχοι που τους συμμεριζόμαστε δεν έχουν επιτευχθεί καθόλου. Τα προβλήματα όμως που αντιμετωπίζουμε έχουν μεγεθυνθεί ακόμα περισσότερο και δεν έχουν καθόλου φυσικά επιλυθεί. Και έχουμε τα προβλήματα της διακυβερνητικής συνεργασίας και εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πώς να το πω, στο τέλος τέλος μπορούμε να θέσουμε και πρέπει να θέσουμε τον δάκτυλο επί του τύπου των ύλων. Και είναι σημαντικό να το κάνουμε για να βρούμε λύσεις, προσεγγίσεις για την επίλυση των προβλημάτων και όλοι οι εμπλεκόμενοι να κινηθούν και να κινητοποιηθούν επικοδομητικά να προχωρήσουν αυτή τη διαδικασία προς τα εμπρός και να σημειωθεί πρόοδος. Ένα από τα σημεία που μας κινεί περισσότερο ως Κοινοβούλιο και εμένα με κινεί είναι το θέμα της κινητικότητας των φοιτητών. Έχουμε αυτό το υπέροχο πρόγραμμα Έρασμος. Όλοι είμαστε τόσο υπερήφανοι και δίκαια γι' αυτό. Είναι ένα καλό πρόγραμμα αυτό και είναι πραγματικά ένα συμβολικό, εμβληματικό πρόγραμμα για την Ευρώπη. Με τη διαδικασία της Μπολόνια, διαδικασίες του έρασμου λιγότερο χρησιμοποιούνται, ακόμα λιγότερο από ό,τι στο παρελθόν. Όταν ακούω από τη Γερμανία και υπάρχουν μελέτες σχετικά ότι σήμερα με τα νέα μαθήματα επιπτυχίο, με τα πτυχιακά, μάστερ, πάρα πολλοί φοιτητέ ε, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να μπορούν να πηγαίνουν στο εξωτερικό ενώ παλαιότερα ε, ήταν 23% αυτό το ποσοστό και σήμερα έχει συρρυκνωθεί. Κάτι δεν πάει καλά λοιπόν. Και πρόκειται για την αναγνώριση σπουδών. Λέει ο Έρασμος, αυτά που έχουν γίνει και τα μαθήματα και τα πιστοποιητικά που έχουν αποκτηθεί στην Αλοδαπή πρέπει και στην Ήμεδαπή, στη χώρα τους, να, είναι, να αναγνωρίζονται. Βλέπουμε αυτά που κάνουν όμως οι φοιτές στο εξωτερικό δεν αναγνωρίζονται στις χώρες τους. Όταν λέμε τα πτυχία πρέπει πανευρωπαϊκά να, είναι, να αναγνωρίζονται, λογικός ο στόχος πανευρωπαϊκά. Όταν διαπιστώνουμε ότι η αλλαγή ενός πανεπιστημίου σε ένα κράτος μέλος το ίδιο, στη Γερμανία για παράδειγμα, δεν είναι δυνατόν επειδή έχουν τόσο εξειδικευτεί τα πανεπιστήμια στα μαθήματα που προσφέρουν, ώστε δεν είναι δυνατόν το Πανεπιστήμιο του Μίνστερ να αναγνωρίζει πιστοποιητικά του Βούπερταλ ε τότε κάτι δεν πάει καλά, κάτι πάει πολύ στραβά και πόρο απέχουμε από αυτά που θα έπρεπε να πετύχουμε με τη διαδικασία της Μπολόνια. Και γι' αυτό είναι σημαντικό και λογικό να ασχοληθούμε με αυτή την έκθεση και να δούμε όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία προανέφερα, γιατί υπάρχουν και πολλά περισσότερα και που ο κύριος Μπερλιγκουέρ ανέφερε στην εισήγησή του Πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας σε αυτά τα θέματα, ελπίζοντας ότι θα μπορέσουμε με τις συζητήσεις που θα κάνουμε να κινητοποιήσουμε τα πράγματα, να κινήσουμε τα πράγματα στην Ευρώπη και με τη διακυβερνητική συνεργασία να πάμε πιο πέρα από ότι τα τελευταία χρόνια. Αυτό που πετύχαμε μέχρι σήμερα είναι ολέθριο. Δεν είναι καθόλου θετικό. Ευχαριστώ. παρακαλώ. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με όλα όσα μας παρουσίασε ο κύριος Μπερλίνγκουερ και αυτό μας ενδιαφέρει δεν είναι μόνο η εθνική οπτική γωνία. Η αναγνώριση των ακαδημαϊκών τίτλων θα πρέπει να γίνει κατά τον πλέον αυτόματο τρόπο Κατά παράδοξο τρόπο, οι τίτλοι οι οποίοι αναγνωρίζονται πιο εύκολα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Υπήρου ή διεθνώς είναι τα διπλώματα, επιστημονικά διπλώματα, δηλαδή των θετικών επιστημών. Εγώ προέρχομαι από ανθρωπιστικές καθαρά σπουδές και νομίζω ότι μεγαλύτερη ε, δυσκολία έγκυται τους ε, στις ανθρωπιστικές επιστήμες, γιατί τα μαθηματικά είναι μία ενιαία παγκοσμίω γλώσσα, αλλά όποιος έχει ένα δίπλωμα ε, φιλολογίας ή ιταλικών σπουδών ιταλικής γλώσσας, είναι δύσκολο να τύχει αναγνώριση αλλού. Αυτό αφορά λοιπόν τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Θα πρέπει λοιπόν να υπογραμμιστεί στην έκθεση αυτή Ε, εδώ φαίνεται ότι δεν είμαι τεχνικός, τεχνικής προσέγγισης, έσβησε το μικρόφωνο μου και δεν το πήρα είδηση. περιπτώσει, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να δεχτούμε ορισμένες επικρίσεις που δεν προέρχονται από καθαρά επιστημονικής, τεχνικής προσέγγισης ε, τύπους και προελεύσεων. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει θα, έπρεπε να ανταγωνιστούμε τους τεχνικούς, τους μαθηματικούς, τις ε, θετικές επιστήμες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τους Κινέζους και τους Ινδούς. Αλλά δυστυχώς οι ανθρωπιστικές επιστήμες φαίνουν ε, στην άκρη γιατί όταν μιλάμε για ανθρωπιστικές ε, σπουδές, ε, όταν οι φοιτητές ε, πηγαίνουν ανά τον κόσμο και ταξιδεύουν για να μάθουν ή να εκπαιδευτούν στην φιλολογία, στην λογοτεχνία, ας πούμε, της Ισπανίας, πήγαιναν από την Ιταλία στην Ισπανία, το έκαναν αυτό επειδή τους άρεσε, επειδή τους ευχαριστούσε. Υπήρχε λοιπόν μια ένα, ενός τύπου καθολικότητα στην Ευρώπη ως προς τις σπουδέ αυτές. Γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να μιλήσουμε για ενοποίηση αναγνώρισης τίτλων, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και όλες αυτές τις πτυχές που είναι καθαρά εκπαιδευτικής προσέγγισης ως προς την, ε, τον διεθνή αυτό χαρακτήρα των τίτλων. Ένα από τα ζητήματα που μας απασχολούν και όπου υπάρχουν ελλείψεις ή κενά είναι από τα πανεπιστήμια τα οποία ανθίστανται στη διαδικασία της ε, Μπολόνια. Μιλάμε δηλαδή για ένα αγγλοσαξονικό πρότυπο. Δηλαδή ένας καθηγητής τακτικός καθηγητής ε, της φιλοσοφικής ο οποίος θέλει να αποκτήσει μία έδρα θα πρέπει να δημοσιεύσει στα αγγλικά, διότι ζούμε σε έναν αγγλοκεντρικό κόσμο. Γιατί πια τα αγγλικά που ισχύουν ως lingua franca δεν είναι αγγλικά, είναι ένα είδος εσπεράντο. Γι' αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις απαιτήσει και τις προαπαιτήσει έτσι ώστε να λάβουμε υπόψη την πολυεδρικότητα των ευρωπαϊκών σπουδών, ιδιαίτερα όσο αφορά τις ανθρωπιστικές σπουδές. Δεν βρήκα κάποια λύση, απλώς θα ήθελα ο συνάδελφος Μπερλιγκουέρ να λάβει υπόψη και αυτή την πτυχή του θέματος, γιατί Μιλάμε για ένα πανεπιστήμιο ευρωπαϊκής εμβέλειας που δεν θα πρέπει να επανεφεύρουμε. Δηλαδή η αναγνώριση πτυχίων βασίζεται περισσότερο στις ε, θετικές επιστήμες, δηλαδή οι ιατρικές σπουδέ είναι ίδιες παντού. Όλες, όλοι πρέπει να γνωρίζουν πώς λειτουργεί το κεντρικό νευρικό σύστημα, πώς έχει η, κυκλοφορία του αίματος, πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος οργανισμός. Εκεί υπάρχει καθολικός χαρακτήρας, αλλά μιλάμε για απαιτήσει που δεν ξέρουμε πώς μπορούμε να ικανοποιήσουμε όταν πρόκειται για ανθρωπιστικές σπουδέ, όπου δεν υπάρχει αυτή η καθολικότητα. Επίσης, αυτό που μας απασχολεί στα μεμονωμένα πανεπιστήμια είναι ο πολυσχηδής χαρακτήρας της γραφειοκρατίας που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε, ιδιαίτερα όταν θα θέλαμε να μεταβούμε κάπου αλλού. Αυτό αφορά και το επίπεδο των περιφερειών και μέσα στην Ιταλία. Όταν κανείς ζητά μία επιδότηση θα πρέπει να διαθέτει γνώση σε ευρωπαϊκού επίπεδου, δηλαδή να υπάρχει ένα γραφείο το οποίο να τον διευκολύνει σε επίπεδο ευρωπαϊκών σπουδών και ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. Θα πρέπει να υπάρχει ένα είδος μεσητείας δηλαδή. Το ίδιο ισχύει και για τις ευρωπαϊκές διαδικασίες. Ίσως θα πρέπει να ε, απλουστευτούν, να απλουστευτεί αυτή η γραφειοκρατία σε συλλογικό επίπεδο. Επίσης κάτι άλλο που με απασχολεί είναι η διαφορά αναγνώρισης τίτλων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτό ε, αφορά και τις συνθήκες σπουδών με μία Ισπανή, Ισπανίδα συνάδελφο σε μία προγενέστερη θητεία μου προσπάθησα να ε, βρούμε, προσπαθήσαμε να βρούμε παραμέτρους τύπου Μάστριχτ για τα πανεπιστήμια. Υπάρχουν πανεπιστήμια στην Ιταλία και αλλού όπου η σχέση διδακτικού προσωπικού και φοιτητών είναι ελιπέστατη. Δηλαδή υπάρχει μια ποσοστή αναλογία διδακτικού προσωπικού σε σχέση με τους φοιτητές όπου δεν υπάρχουν συγκεκριμένα εχέγγυα σπουδών, δηλαδή δεν υπάρχουν αρκετές βιβλιοθήκες, δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχουν αρκετές υποτροφίες. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν βασικά κριτήρια διευκόλυνσης και προσβασιμότητας δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα μπορούσε να ενταχθεί στην έκθεση του κυρίου Μπερλιγκουέρ, αλλά θα έπρεπε κατά κάποιο τρόπο να βρεθεί μία λύση. Διότι και στις χώρες της Μεσογειακής Λεκάνης, με τις μεταναστευτικές ροές, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τα πανεπιστήμια από τις χώρες του Μαγκρέμπ, της Βορείου Αφρικής. Διότι Αυτές οι μεταναστευτικές ροές αλλάζουν και τα πολιτισμικά δεδομένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Εκτός μικροφώνου κυρία Σήμερα δεν μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα όλων των πανεπιστημίων. Μιλάμε για την Πολόνια. Όλα όσα είπατε είναι σωστά. Πρέπει όμως κάπως να περιοριστούμε στο ουσιαστικό μας θέμα. Είναι μια Ιταλο-Ιταλική συζήτηση αυτή. Κυρία Κώστα, παρακαλώ. Θα ήθελα να πω ε, χαίρομαι που βρίσκομαι μαζί με Ιταλούς και συζητάω, ένα πολύ ενδιαφέρον. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Λουίτζι Μπελιγκουέρ, ε, διότι όχι μόνο για αυτή την έκθεση που είναι τόσο θαραλέα και τόσο ε, σαφής ε, αλλά και για το πάθος που μας εμπνέει και για την ε, προσωπική και πολιτική θα έλεγα αξιοπιστία με την οποία εδώ και καιρό αυτός ο ίδιος που στηρίζει αυτή τη διαδικασία και παρέχει κίνητρα σε όλους τους παράγοντες σε εθνικό επίπεδο και στο ευρωπαϊκό επίπεδο και βοηθάει να προχωρήσουν τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Μου φαίνεται ότι αυτή η έκθεση έχει τη φιλοδοξία και εν ώψη της επόμενης ε, διάσκεψης των Υπουργών το 2012 να πάμε πιο πέρα από το θέμα της πρόθεσης της κινητικότητας των ε, φοιτητών ε, που υπάρχουν στο πλαίσιο του Εράσμους και που φυσικά υπήρξε ένα θεμελιώδη στοιχείο αλλά το να μπούμε στην καρδιά ουσιαστικά της διαδικασίας της Μπολόνια χρειάζεται τεράστιο θάρρος ώστε να αξιολογήσουμε σωστά το ζήτημα της επικουρικότητας το οποίο δεν θα πρέπει να αποτελέσει δικαιολογία για να για να διασφαλίσουμε το δικαίωμα των νέων αλλά και στο οι οποίοι πρόκειται να απασχοληθούν στο μέλλον. Δεν θα, θα πρέπει λοιπόν να τους ενθαρρύνουμε να μπορούν να σπουδάσουν, να ακολουθήσουν την ακαδημαϊκή τους πορεία σε οποιοδήποτε ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο υπό τις κατάλληλες συνθήκες. Αυτές μου, αυτή μου φαίνεται ότι είναι ο στρατηγικός στόχος από τον οποίο, στον οποίο βασίζεται η διαδικασία της Μπολόνια. Όλες οι δράσεις που μπορούν να μας οδηγήσουν προς αυτή την κατεύθυνση στο πλαίσιο φυσικά της νομικής βάσης που μας παρέχει η Λισαβόνα ε, για τη δυνατότητα μεταφοράς και αμοιβέ αναγνώρισης των τίτλων πιστεύω ότι εδώ νομιμοποιείται μια νέα πιο θαραλέα φάση που θα πρέπει να ακολουθήσουμε ε, συμφωνώ με τους ε, ενδιασμούς που ακούστηκαν και τις ανησυχίες καταλαβαίνω και το βλέπω, γνωρίζουμε πώς πάνε τα πράγματα, ότι η αναγνώριση ακαδημαϊκών μονάδων και τίτλων στον τομέα των ανθρωπιστικών σπουδών ε, είναι πιο περιπλοκή από τον επιστημονικό τομέα. Ωστόσο η πρόταση που γίνεται στην έκθεση του κυρίου Μπερλιγκουέρ είναι να καταφέρουμε να καθορίσουμε κάποιο πυρήνα κατά κάποιο τρόπο που θα μπορεί να αποτελέσει ένα σημείο αμοιβαίας αναγνώρισης και το οποίο θα ε, σέβεται τις πολιτισμικές διαφορές και τις διάφορες, ε, διαφορετικές διαδικα... διδακτικές διαδικασίες. Ιστορικά η διαδικασία της Μπολόνια δημιουργήθηκε από, τις, από τα κράτη-μέλη, από τις κυβερνήσεις, αποτέλεσε μετά αντικείμενο των Πριτάνων και μετά αποτέλεσε μια νέα διδακτική στρατηγική μεταξύ του διδακτικού προσωπικού και αποτελεί ένα νέο στοιχείο ηθαγένειας μεταξύ των φοιτητών. Θα θέλουμε λοιπόν να υπάρχει δυνατότητα να δημιουργήσει κάποιο το δικό του πρόγραμμα σπουδών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ήθελα απλά να υπογραμμίσω ότι υποστηρίζουμε και τη μεθοδολογία, τη διακυβέρνηση, τα εμπόδια, τα σημεία συμφόρηση και τις δράσεις που πρέπει να αναλάβει η Ευρώπη. Θα ήθελα να προσθεθεί ότι το όσον αφορά το δικαίωμα σπουδών έχουμε ευρωπαϊκά δίκτυα πολύ σημαντικά και εθνικά ή περιφερειακά ιδρύματα που παρέχουν το δικαίωμα ε, σπουδών. Μιλάω για τις υποτροφίες, για βιβλιοθήκες, εργαστήρια, όλα αυτά που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της πραγματικής ευκαιρίας που προσφέρεται στα παιδιά να αισθανθούν ότι είναι Ευρωπαίοι πολίτες. Όλοι αυτοί οι παράγοντες ζητούν τη φορητότητα των διαφόρων παροχών, της πρόσβασης ας πούμε στη, σε κατοικία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κατά την άποψή μου αυτό το κομμάτι έχει παραβλεφθεί κατά κάποιο τρόπο ενώ αποτελεί θεμελιώδες ε, στοιχείο και υπάρχουν και σχετικές εκθέσεις. Στην Ιταλία, το δεύτερο που ήθελα να πω σήμερα και το υπογράμμισε ο κύριος Μπερλιγκουέρ, έγινε μια πολύ σημαντική συμφωνία μεταξύ της Confindustria και των Λυκείων για το ζήτημα του διδακτορικού έρευνας σε επιχειρήσεις. Επειδή η κυρία Βασιλείου ανακοίνωσε ότι θέλει να δημιουργήσει μία νέα κινητικότητα στα μάστερ, εγώ θα πρότεινα αυτό το θέμα να συμπεριληφθεί σε αυτή τη δυνατότητα των μάστερ σε συμφωνία όχι μόνο με τις επιχειρήσεις αλλά, με και, τους φορείς που, αλλά και με τους φορείς που απασχολούνται με άλλους ε, τομείς όπως με την αρχαιολογία. Ένα τελευταίο πράγμα που ήθελα να πω, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το μείγμα και η ομογενοποίηση που πολλές φορές δεν καταφέρνουμε να επιτύχουμε ε, και που δεν θέλουμε ίσως γιατί δεν θέλουμε ευρωπαϊκό πρόγραμμα σπουδών αυτή, αυτή, αυτός ο συνδυασμός μεταξύ της εμπιστοσύνης θεμελιώδου στοιχείου του περιεχομένου αυτού του πυρήνα ε, εκπαίδευσης και τα συστήματα διασφάλισης της ποιότητας. Σε αυτούς τους τομείς η Ευρώπη μπορεί να κάνει περισσότερα. Πιστεύω ότι η Ευρώπη ε, υιοθετώντα ε, στα συστήματα αξιολόγησης των πανεπιστημίων τη δυνατότητα προώθησης της κινητικότητας όχι μόνο των φοιτητών αλλά και του διδακτικού προσωπικού αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μια παράμετρο που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και στους διαφόρους δείκτες που, στους οποίους βασιζόμαστε για, τις, ε, για, την, για την παρακολούθηση της πορείας του όλου πράγματος. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Παλιατέλη παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, ομολογώ ότι θα πρέπει να ευχαριστήσω τον κύριο Μπερλίνγκορ και για έναν ακόμη λόγο πέρα από αυτούς που υπόθηκαν ε, από τους ε, προλαλήσαντες γιατί η πρόταση για την έκθεση, η έκθεση του αυτή έρχεται σε μια ε, είναι πολύ επίκαιρη για μια ε, διαδικασία που ε, νομιμοποιήθηκε δέκα χρόνια πριν σε μια άλλη Ευρώπη και που έρχεται να αποτιμηθεί δέκα χρόνια αργότερα σε μια νέα Ευρώπη. Από αυτή την άποψη θεωρώ ότι είναι ακρούς πολιτική η προσέγγιση του καθηγητή Μπερλίνγκουερ στην παιδεία, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση γιατί κατά βάση περιγράφει και αντανακλά ζητήματα που αντιμετωπίζουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, η έκθεση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα βαθμό σαν εργαλείο για να κρούσουμε τον κόδωνα του κινδύνου σε μια Ευρώπη ε, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο να μην συνεχίσει αυτή που ήταν ε, λίγα, χρόνια πριν. Ε, θεωρώ επομένως πολύτιμη αυτή την ε, έκθεση και χαίρομαι ότι, οι ότι δεν είμαι μόνη σε αυτό το χώρο σε ό,τι αφορά τις ανθρωπιστικές τις οποίες αντιλαμβάνομαι περισσότερο όχι ως ε, προσπάθεια αυτών που τις διδάσκουν για αυτούς που τις διδάσκουν για την ε, επαγγελματική τους αποκατάσταση και μόνο αλλά ως εργαλείο για ένα νέο μοντέλο Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου στο οποίο οι ανθρωπιστικές σπουδές παίζουν κέριο ρόλο ως αντίβαρο σε ένα μοντέλο πανεπιστημίων αγγλοσαξονικού τύπου που μας οδήγησαν ενδεχομένως και στην οικονομική κρίση την οποία βιώνουμε αυτή τη στιγμή ακριβώς επειδή λείπει μια ευρύτερη παιδεία από την πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Φοβάμαι ότι τα golden boys της εποχής μας δεν έχουν ακούσει τις ανθρωπιστικές σπουδέ ή δεν τις έχουν εστερνιστεί Θεωρώ, για θα είμαι πολύ σύντομη, ότι η αξιολόγηση είναι το υπαριθμόν ένα προϋπόθεση για την εγκυρότητα κάθε κύκλου. Άρα η αξιολόγηση πρέπει να αποχωρήσει σε όλες τις χώρες προκειμένου να προκύψει στη συνέχεια μια γενικότερη ευρωπαϊκή αξιολόγηση. Και όλες οι χώρες νομίζω ότι πρέπει να αποδεχτούν ως δεύτερη προϋπόθεση την τριμερή δομή, δηλαδή το bachelor, την τριετή φίτηση, το μάστερ και το, και διδακτορικό ε, κύκλο. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να τα επιβάλλουμε σχεδόν υπερβαίνοντας ε, το πρόβλημα της ε, επικουρικότητας με το επιχείρημα ότι είναι εργαλεία και πάλι για την, όχι για την κινητικότητα μόνο αλλά και για την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφύτων των πανεπιστημίων και αυτό η employability, η ε, ε, αποσχολησιμότητα αφορά την, Ευρώπη, ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι θέμα επικουρικότητας. Αφορά το μέλλον της Ευρώπης, το νέο σε επαγγελματικό επίπεδο. Πρέπει επίσης νομίζω να προσπαθήσουμε να συντονίσουμε τις, τους διάφορους οργανισμούς που ασχολούνται με την ευρωπαϊκή τριτοβάθμια εκπαίδευση με έναν τρόπο που θα είναι πιο ευανάγνωστοι. Δηλαδή, η ευρωπαϊκή ε, ε, ε, ευρωπαϊκή European Higher Education Area και η European Research Area θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να συντονίζονται. Ακόμη και σε ό,τι αφορά τα προγράμματα, τα ερευνητικά που ε, κατατίθενται από την Επιτροπή. Και δεν καταλαβαίνω τον ρόλο πώς πώς συνεργάζεται το European Union Association με αυτούς τους δύο βασικούς ε, ε, άλλους φορείς. Εκτιμώ λοιπόν ότι πρέπει να απλοποιήσουμε, να, να συγκροτήσουμε έναν πυρήνα που θα περιλαμβάνει όλους αυτούς τους επιμέρους οργανισμούς και επομένως θα εγγυάται το ότι θα συντονίζει σε έναν βαθμό αυτά που είπα λίγο πριν. Θεωρώ όμως τελικά, και τελειώνω εδώ κυρία Πρόεδρε, ως εξαιρετικά επίγον να βρεθεί ένας τρόπος αξιολόγησης των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και κατάταξής τους όχι με βάση τα κριτήρια των διάφορων τη Σανγκάη, του δεν ξέρω τι, όπου οι ανθρωπιστικές σπουδές και άλλα, και άλλα πράγματα δεν παίζουν κανένα ρόλο. Πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά επίγον να συσταθεί ένα σύστημα ευρωπαϊκό για την αξιολόγηση στην οποία θα περιλαμβάνονται και η εμπειρία μας στην εκπαίδευση και αυτό ίσως αποτελέσει μοχλό για το να γίνουν τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια περισσότερο ελκυστικά για τους ε, μη Ευρωπαίους πολίτες. Επομένως είναι κατεπήγον για μένα να αντισταθούμε με ένα νέο τρόπο και με νέα κριτήρια σε αυτή την πολύ επιδερμική ε, προσέγγιση για την, για την κατάταξη των πανεπιστημίων του κόσμου με βάση κριτήρια που δεν ανταποκρίνονται ε, σε αξίες αλλά μόνο σε αριθμούς. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Παλιαδέλη. Με την αξιολόγηση των σχολείων πρέπει κάπως, των πανεπιστημίων να είμαστε κάπως ε, προσεκτικοί. Πρέπει να είμαστε κάπως πιο επιφυλακτικοί. Δεν θέλουμε ranking και αυτό το είπαμε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ξέρουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει κάτι τελείω ε, διαφορετικό και πρέπει αυτό να, είναι, να το θεωρούμε καλό και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στην αξιολόγηση. Δεν θέλω να σα διορθώσω, δεν θέλω τίποτα να διορθώσω, αλλά πρέπει να ξέρουμε ακριβώ τι θέλουμε, τι επιθυμούμε. Ότι δεν θέλουμε ranking το γνωρίζουμε, αλλά μια αξιολόγηση όπω το κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε, με διαφορετικές προσφορές, ας το πω έτσι, κύκλων σπουδών, ότι μπορεί να δεχθεί έτσι να, στους υποψήφιους πώς μπορούν να σπουδάσουν καλύτερα το ένα ή άλλο αντικείμενο, γνωστικό αντικείμενο. Ranking όμως δεν θέλουμε. Δεν ήταν αυτό το οποίο εννοούσες, έτσι δεν είναι. Θα επανέλθουμε στη συνέχεια σε αυτό. Ωραία, εντάξει. yes, But with new criteria. Ah, Εντάξει, το εννοούσατε με νέα κριτήρια. Εντάξει, ενδιαφέρον. Δεν είναι πάντα το ίδιο το ranking όταν μιλάμε για ένα αντικείμενο. Κύριε Σκουρία, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν είχαμε καμία αμφιβολία ότι ο κύριος Μπερλιγκουέρ θα ήξερε να προσεγγίσει το θέμα υπό τη σωστή οπτική γωνία, ότι θα είχε τη σωστή προσέγγιση. Θα ήθελα όμως να υποστηρίξω δύο πτυχές. Πρόκειται για δυσεπίλητα θέματα. Καταρχήν ως προς τους τίτλους σπουδών και την εναρμόνιση υπό την έννοια της προσέγγισης της αγοράς εργασίας. Σήμερα στην Ευρώπη μας έχουμε πολλές διαφορές πολύ μεγάλες διαφορές, έτσι ώστε όταν ένας φοιτητής τελειώνει τις σπουδές του στην Ισπανία, ας πούμε, και θέλει να ασκήσει το επάγγελμα του δικηγόρου, βλέπει ότι σε άλλες χώρες υπάρχουν διαφορετικές προσέγγισεις και διαφορετικά εχέγγυα σε μια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η εναρμόνιση λοιπόν είναι θεμελιώδους σημασίας εάν θέλουμε μια κοινή αγορά εργασίας. Θα πρέπει όμως στην αγορά εργασίας να μπορούν να εισέλθουν άνθρωποι που έχουν τους ίδιους τίτλους σπουδών, με το ίδιο περιεχόμενο δηλαδή σπουδών. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μία μεγάλη απειλή και θα πρέπει να μας απασχολήσει. Υπάρχουν πολλά πανεπιστήμια όπου για να μπορέσει να μπει κανείς υπάρχει ο κλειστός αριθμός, το νούμερο κλάουζους, σύμφωνα με το οποίο μπορεί κανείς να μπει όχι σε ένα πανεπιστήμιο. Επειδή λοιπόν υπάρχει ο κλειστός αριθμός, δεν μπόρεσαν να σπουδάσουν πολλά παιδιά, πολλοί φοιτητέ και μέσα στα πλαίσια της κινητικότητας φοιτητέ μεταφέρονται σε άλλα πανεπιστήμια τα οποία έναντι αντιτίμου εγγράφονται στα πανεπιστήμια και το δεύτερο χρόνο, τη δεύτερη χρονιά σπουδών προσπαθούν να ξαναμπούν στη χώρα υποδοχής, στο πανεπιστήμιο ε, της χώρας υποδοχής, όπου δεν μπόρεσαν να εισέλθουν καταρχήν. Ενώ άλλοι φοιτητέ με υψηλότερη βαθμολογία μπόρεσαν να μπουν εξ αρχής έτσι ώστε να υπάρχει και ένα συγκεκριμένο επίπεδο ε, σπουδών. Και αυτό νομίζω ότι δεν ε, υπεραμείνεται της έννοιας της κινητικότητας γιατί εδώ υπάρχει μία εντελώς ε, διαφορετική τελεολογία η οποία δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από εμάς. Πρόκειται για ένα νέο φαινόμενο, το οποίο όμως προσλαμβάνει διαστάσεις και θα ήθελα ο κύριος Μπερλουγκουέρ να ασχοληθεί και με αυτή την πτυχή του ζητήματος, έτσι ώστε να λάβει υπόψη και αυτή την ε, πλευρά της μεταφοράς, της δυνατότητας μεταφοράς, ε, κάτω από αυτούς τους όρους. Σας ευχαριστούμε κύριε Βενέρα Πατού παρακαλώ. Euh, ναι, ευχαριστούμε κύριε Μπερλιγκουέρ για αυτή τη γενική εικόνα, αυτό το πανόραμα που μας περιγράψατε. Ε, μία ερώτηση πρώτα απ' όλα που αφορά το καθεστώς των φοιτητών στη Γαλλία στο πρώτο έτος του Πανεπιστημίου. Το πρώτο έτος του Πανεπιστημίου είναι έτος προσανατολισμού. Υπάρχει μεγάλο ποσοστό αποτυχιών. Επίσης υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα ότι σε κοινωνικό επίπεδο πολύ λίγοι ε, φοιτητέ προέρχονται από τα λαϊκά στρώματα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Συχνά επίσης ε, δεδομένου του ποσοστού της ανεργίας στο πανεπιστήμιο και ειδικότερα το πρώτο έτος ε, είναι ένας τρόπος να έχει κάποιος κάποιο καθεστώς όταν δεν έχει δουλειά. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε Ποιο είναι ο συνδέσμος μεταξύ της διαδικασίας της Μπολόνια και των τεχνολογικών διπλωμάτων. Στη Γαλλία τα επαγγελματικής κατάρτισης ε, η τεχνολογικά ε, είναι, είναι ένα ε, στύπου, είναι ένα τύπου απολυτήριο με το οποίο δεν επιτρέπει να πάει στο πανεπιστήμιο κάποιος. Ε, για να υπάρχει λοιπόν διαβίου εκπαίδευση θα πρέπει να μπορεί να μπει κάποιο και να βγει από το πανεπιστήμιο. Μου φαίνεται ότι είναι σημαντικό το πανεπιστήμιο να είναι πιο ανοιχτό, να επιτρέπει και την είσοδο και την έξοδο ε, και όχι να μπαίνει κάποιο να ακολουθεί όλη τη διαδικασία και να μην μπορεί να ε, πάρει πτυχίο. Επίσης υπάρχουν όλο και περισσότερα τα πανεπιστήμια τρίτης ηλικίας, όλο και περισσότεροι άνθρωποι που σε μεγάλη ηλικία θέλουν να ε, σπουδάσουν αυτό συνήθω δεν συμβαίνει μέσα στο πανεπιστήμιο, μέσα στο πανεπιστημιακό χώρο αλλά δίπλα. Θα πρέπει λοιπόν τα πανεπιστήμια να είναι πιο ανοιχτά προ την κοινωνία, να δίνουν τη δυνατότητα στου φοιτητέ από τα λαϊκά στρώματα να εισέρχονται, να υπάρξει κάποια σύνδεση με τα τεχνολογικά πολιτήρια, τα τεχνολογικά διπλώματα και τα επαγγελματικά διπλώματα. Τέλο όσον αφορά τις δημοσιεύσεις ε, για να, γίνει να υπάρχει μια σχέση με τον τομέα της έρευνας, το είπατε και εσείς, είναι πολύ σημαντικό η έρευνα να μπορέσει να σχετιστεί με τα πανεπιστήμια. Μιλήσατε για τις ανθρωπιστικές επιστήμες, συμφωνώ απόλυτα. Είναι ένας πολύπλοκος τομέας και οι ανθρωπιστικές επιστήμες ε, πρέπει να περιλαμβάνονται όχι μόνο με στα προγράμματα σπουδών, αλλά και στις ε, επιστημονικές ε, σπουδές, να υπάρχουν κριτικές φιλοσοφικές προσεγγίσεις ε, και στην ιατρική κτλ. Πιστεύω ότι θα πρέπει να μπορέσουμε να συζητήσουμε για τι δημοσιεύσεις. Οι περισσότερε δημοσιεύσει σήμερα είναι στα αγγλικά και έχουμε μία αγγλοσαξονική προσέγγιση ως επιτοπλίστων. Θα πρέπει ως Ευρωπαίοι να μπορέσουμε να αναπτύξουμε και να υποστηρίξουμε ευρωπαϊκές δημοσιεύσει με τις ε, διαφορετικότητες των γλωσσών στα γαλλικά, στα ιταλικά Μιλήσαμε προηγουμένως, ο κύριος Μάτιμο μίλησε για τη Μεσόγειο, εσείς μιλήσατε για 47 χώρες, πολλές χώρες του Νότου έχουν υλοποιήσει αυτή τη διαδικασία της Μπολόνια. Υπάρχει ένα ρουμάνικο πανεπιστήμιο το οποίο έχει ανταλλαγές τώρα με τη Σλοβενία. Υπάρχει μια ομάδα εργασίας στο Ρουμανικό Κοινοβουλίο. Υπάρχει ένα δεύτερο πανεπιστήμιο ε, Ευρώπης και Μεσογείου θα δημιουργηθεί στο ΦΕΣ στο Μαρόκο και πολλές χώρες θα θέλαν ένα Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και σε άλλα μέρη του Νότου. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει δυνατότητα συγκρίσεων με άλλα προγράμματα σπουδών. Έχουμε πολλές αναδυόμενες οικονομίες στην Κίνα, τη Βραζιλία, την Νοτιοφρική, τη Ρωσία θα καλό θα ήταν να μάθουμε τι προγράμματα υπάρχουν σε αυτές τις χώρες, πώς ένας Ευρωπαίος θα μπορούσε ενδεχομένω να ενσωματώσει ή να αναγνωρίσει ένα βραζιλιάνικο ή ινδικό πτυχίο. Ε, Τελευταίος εξίσου σημαντικός, η κυρία Χάνιμπαλ, παρακαλώ. Um, Ευχαριστώ. Στα αγγλικά μια παρέμβαση, μια και έχουμε και το θέμα των αγγλικών σε αυτή τη συζήτηση κάποια πράγματα υπό τους διαφορετικούς τίτλους ε, κατηγορίες θα ήθελα να πω. Να ευχαριστήσω πρώτα τον κύριο Μπέρλινγκουε Πολύ ενδιαφέρουσα και δυναμική συζήτηση. Μια καλή βάση, καλά θεμέλια να προχωρήσει αυτή η έκθεση και να προαχθεί το θέμα. Το πρώτο που θα ήθελα να αναφέρω είναι η αυτονομία των πανεπιστημίων, πανεπιστημιακών ιδρυμάτων θα έπρεπε να δούμε μια ευρωπαϊκή πτυχή και κινητικότητα. Ένα από τα θέματα που στην Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή κάνουμε πολύ συχνά λόγο είναι ακριβώς η αυτονομία. Πρέπει τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, ακαδημαϊκά ιδρύματα σε αυτό το επίπεδο να μπορούν να συναποφασίζουν σε μεγάλο βαθμό πώς θα διοργανώνουν τα μαθήματα που προσφέρουν και πώς θα το κάνουν και ε, όταν έχουμε το θέμα των υψηλών προδιαγραφών και στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Αυτό που επιλέγουν να διδάσκουν τα πανεπιστήμια είναι εκείνο στο οποίο θα πρέπει να αποφασίζουν αυτοτελώς και αυτοβούλος, με αυτονομία. Και πιστεύω ότι ακριβώς μέρος ε, από το ε, πανεπιστημιακό φάσμα, σημαντικό τμήμα, είναι η ποικιλότητα, η πολυμορφία και πολυσχεδής τρόπος προσφορών μαθημάτων να μπορούν να είναι και ανοιχτά και διαφανή αυτά όλα. Μέρος του προβλήματος είναι ότι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν και να διαδώσουν προς τα έξω αυτό το οποίο κάνουν τα πανεπιστήμια. Υπάρχει έλλειψη γνώσεων για το τι τεκταίνεται στα πανεπιστήμια. Κάποιο σύστημα αξιολόγησης λοιπόν, καθώς επίσης και η διασφάλιση ότι τα ίδια τα, τα, ίδια πανεπιστήμια θα γνωστοποιούν προς τα έξω το τι κάνουν, ώστε να γνωρίζουν οι άλλοι ότι προσφέρεται το ένα ή άλλο μάθημα, αυτό νομίζω πολλά θα διευθετούσε και θα επέτρεπε την ποικιλότητα και τον πολυσχηδή χαρακτήρα των μαθημάτων στις ανθρωπιστικές σπουδές. Δεν ξέρω τι γίνεται με τις διαφορετικές χώρες, αλλά έτσι λειτουργούν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι δική τους δουλειά σε μεγάλο βαθμό με την αυτονομία και αυτοδυναμία που έχουν να λειτουργούν έτσι αυτόνομα. Κι εγώ σπούδασα και ιστορία ουσιαστικά και τα μαθήματα τα, όσα προσφερόντουσαν σε σχέση με την ιστορία στα πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν διαφορετικά μεταξύ τους αλλά πολύ καλό ήταν αυτό. Βρίσκοντας το τι έκαναν μπορούσε ο υποψήφιος πτυχιούχος να αποφασίσει τι θα παρακολουθούσε. Έτσι λειτουργούσαν τα πράγματα. Γιατί να είναι πρόβλημα λοιπόν αυτό τουλάχιστον όσον αφορά τι ανθρωπιστικές σπουδές. Αλλάζουν κάπως τα πράγματα όταν κάνουμε λόγο για επιστήμες θετικές επιστήμες και προσόντα και πτυχία. Υπάρχουν μαθήματα που οδηγούν σε τέτοιου είδους επαγγέλματα όπως στην ιατρική και στα μαθήματα της νομικής επιστήμης στα πτυχία. Να δούμε τι γίνεται ευρωπαϊκά. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα ε, σε γρήγορση και προσεκτικοί και όπως είπε ο κύριος Βάτιμο σε σχέση με την επιστήμη ο τρόπος που λειτουργεί είναι διαφορετικός, είναι πολύ πιο δομημένος και προφανής. Θα μπορούσαμε ίσως να ε, έχουμε κάποιες ε, διαφορετικές απόψεις σε σχέση με την προηγμένη ε, επιστήμη. Λοιπόν, σε σχέση με την επιστήμη, εφαρμοσμένη επιστήμη, καθαρά θεωρητική επιστήμη και επιστήμες που οδηγούν σε επαγγελματικά πτυχία άσκησης επαγγέλματος. Δεν είναι δύσκολο να το δούμε έτσι. Θα διασαφη... πολλά πράγματα σε σχέση με τη συζήτηση. Και εδώ περνάμε τώρα στο ίδιο, το, στην ίδια την προσφορά μαθημάτων στο curriculum. Θα πρέπει να είναι γνωστό ότι διδάσκονται τα α, β, γ μαθήματα και να επαφείτε στα πανεπιστήμια πώς θα το κάνουν αυτό έχοντας συμφωνήσει για τις παραμέτρους της ακαδημαϊκής δραστηριότητας ε, και της ακαδημαϊκής ε, θα έλεγα ε, αριστείας εντός εισαγωγικών έστω και αν αυτό θα μπορούσε να συζητηθεί. Συμφωνώ με την προλαλή σας, πρέπει να δούμε τα θέματα των κοινωνικών επιστημών, να μπορέσουμε να έχουμε τα θέματα τα κοινωνικά. Δεν ξέρω τι γίνεται σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά τα πράγματα έχουν επιδεινωθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πολλά έχουν αναφερθεί για την βελτίωση του, της σύνθεσης των φοιτητών από διάφορα κοινωνικά στρώματα. Ένα από τα πράγματα που θα πρέπει να κάνουμε στα πανεπιστήμια και τα ίδια τα πανεπιστήμια <clears throat> θα πρέπει να είναι αυτό το κοινωνικό μείγμα από διάφορες ε, προελεύσεις και ε, διαστρωματώσεις φοιτητών. Οι περισσότεροι, τουλάχιστον σε σχέση και με τους φοιτητές στα προπτυχιακά, δεν θα φοιτήσουν, δεν θα παρακολουθήσουν κάτι το οποίο θα έχει άμεσα σύνδεση με την επαγγελματική τους δραστηριότητα εκτός αν είναι σε σχέση με τα νομικά, την ιατρική ή κάποιο είδους άλλη επιστήμη. Στο τέλος θα καταλήξουν να ασκήσουν κάποιο επάγγελμα το οποίο δεν θα έχει κάποια άμεση σχέση με τα μαθήματα, τα προπτυχιακά τους. Θα πρέπει να το δούμε αυτό τον διάλογο πανεπιστημίων και επιχειρήσεων ε, κόσμου ε, της, ε, του επιχειρήν πρέπει να το δούμε σε στενή διασύνδεση. Αν θέλουν να το κάνουν αυτό τα πανεπιστήμια και να επεκταθούν σε αυτό θα μπορούσαμε να το επεκτείνουμε περαιτέρω ώστε τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια συνολικά να λαμβάνουν περισσότερο υπόψη την πτυχή της απασχόλησης των φοιτητών τους σε συγκεκριμένα επαγγέλματα μετά την απόκτηση κάποιων πτυχίων. Πολύ καλή δουλειά κάνει ο κύριος Μπερλίνγκουερ. Κατά κάποιο τρόπο εξετάζουμε μέσα από τη διεργασία Μπολόνια το ποιο πρότυπο ακολουθείται και πώς αναφέρθηκε το αγγλοσαξονικό πρότυπο. Όταν αναφερόμαστε σε αγγλοσαξονικό εννοούμε συνήθω και τι, ΗΠΑ όπου υπάρχουν φυσικά και τεράστιε διαφορέ, Είναι το βρετανικό πρότυπο. Είναι το αγγλόφωνο, εν πάση περιπτώσει θα λέγαμε πρότυπο όσον αφορά τι ανώτατε σπουδέ. Και αυτό μα δίνει ένα φάσμα, ένα έρο για να δούμε πώ μπορούν να εξεταστούν τα διάφορα θέματα που αναφέρατε σε τρία επίπεδα. Για τη συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών που μετά το προπτυχιακό τους θα αποχωρήσουν. Άλλοι όμως υπάρχουν και που θα ακολουθήσουν ε, ε, τις σπουδές τους μέχρι και το μεταπτυχιακό και θα ανέβουν και ακόμα παραπάνω εξειδικευόμενοι. Πρέπει να σημειώσουμε πρόοδο προς αυτήν την κατεύθυνση και πάλι ευχαριστώ τον κύριο Μπερλιγκουέρ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Άνταμ Τάισεν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μπερλιγκουέρ για την εισήγηση που μας έδωσε. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση με ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Όπως είπατε κυρία Πρόεδρε, πρόκειται για ένα θέμα για την διαδικασία της Μπολόνια αποκλειστικά και γι' αυτό θα αρκεστώ σε αυτήν. Πιστεύουμε ότι η εξυγχρονισμένη ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πιο διευρυμένη από τη Μπολόνια γιατί υπάρχουν πολλές επικαλύψεις και νομίζω ότι θα ήταν πολύ σημαντικό οι δύο διαδικασίες να συνάδουν, να συμπέσουν έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχυθεί στα πλαίσια της διαδικασίας της Μπολόνια. Όπως ελέγχθη, η διαδικασία της Μπολόνια Ξεκινά από την ιδέα ότι θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη κινητικότητα και συνεργασία των πανεπιστημίων των κρατών μελών. Δηλαδή, μιλάμε για τις αλλαγές που είναι αναγκαίες για να δημιουργηθεί εμπιστοσύνη. Άρα, μιλάμε για αμοιβαία αναγνώριση που είναι ύψης της σημασίας για ποιοτικές σπουδές και βεβαίως θέματα προσβασιμότητας στα πανεπιστήμια. Μιλήσαμε και για την κοινωνική διάσταση. Θα ήθελα να αρκεστώ και να μιλήσω για τις τρεις αυτές πτυχές, διότι έγινε μία υπόδειξη υπό την έννοια ότι η διαδικασία της Μπολόνια είναι καταστροφική. Δεν πιστεύω ότι ισχύει αυτό. Έχει γίνει μεγάλη πρόοδο σε όλους τους τομείς της ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης. Βεβαίως βρισκόμαστε σε μια μεταβατική φάση. Όλα και πολλά μάλλον θα πρέπει να διευκρινιστούν με βάση αυτούς τους κύκλους σπουδών και το σύστημα των credits των ε, πιστοτικών μονάδων που υπάρχουν στα μαθήματα. Ως προς την ποιότητα, επίσης έχει επέλθει πρόοδος. Υπάρχουν agencies ποιοτικού ελέγχου σε πολλές χώρες, ίσως εργάζονται κάπως διαφορετικά, αλλά μαθαίνουν οι μεν από τις δε. Αλλά δεν υπάρχει διασυνοριαχή διοσυναριακή διαπίστευση ελέγχου. Εδώ υπάρχουν πολλές ελλείψεις. Όταν ε, μιλάμε για αμοιβαία αναγνώριση, νομίζω ότι αυτό που έχει σημασία είναι η αναγνώριση για, τους, για καθαρά ακαδημαϊκούς σκοπούς, δηλαδή για περαιτέρω σπουδές σε μια άλλη χώρα και μας είπε ε, μία συνάδελφος από τη Γερμανία ότι υπάρχουν μεγάλες ε, ε, δυσκολίες όταν μιλάμε για αναγνωρίσεις και μεταξύ πόλεων της Γερμανίας, δηλαδή από το Μύνστερ μεταξύ Μύνστερ και Βούπερταλ. Αλλά όταν μιλάμε για τη διασυνοριακή κατάσταση αναγνώρισης, θα πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερο. Υπάρχει η Σύμβαση Αναγνώρισης της Λισαβόνας που έχουν κυρώσει όλα τα κράτη-μέλη σχεδόν αλλά υπάρχουν προβλήματα διότι με μονομένα πανεπιστήμια μπορούν να μην αναγνωρίσουν διπλώματα τη στιγμή που θεωρούν ότι υπάρχει μεγάλη απόσταση περιεχομένου σπουδών. Γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει τα πανεπιστήμια και τα ιδρύματα τα ίδια να ορίσουν εξειδικεύσεις χωρίς να αποτελούν πρόσκομα για την κινητικότητα των σπουδαστών. Όταν μιλάμε για την επαγγελματική προσέγγιση των πανεπιστημιακών τίτλων και υπάρχει και μία οδηγία, κοινοτική οδηγία επί του θέματος, όπως ξέρετε θα ε, αλλάξει κάπως η οδηγία μέχρι το τέλος του έτους, έτσι ώστε να λάβουμε υπόψη τις ανάγκες της αγοράς-εργασίας, καθώς και τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα ανά την Ευρώπη. Νομίζω λοιπόν ότι η Επιτροπή σας θα πρέπει να ασχοληθεί με αυτό το θέμα, καθώς και η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς. Όταν μιλάμε για επαγγελματικά προσόντα, ε, όταν μιλάμε δηλαδή για την ασφάλεια των ασθενών ή άλλων πολιτών στα κράτη-μέλη, όταν μιλάμε για αρχιτέκτονες και ούτω καθεξής, θα πρέπει να υπάρχει υψηλότερη, μια υψηλότερη βαθμίδα εμπιστοσύνης και διασφάλισης. Και γι' αυτό θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το σύστημα ε, πιστοτικών μονάδων και ε, μεταφοράς πιστοτικών μονάδων, μονάδων πίστοση σε άλλα κράτη-μέλη. Θα πρέπει λοιπόν η νέα οδηγία να έχει μια ευελιξία μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας της Μπολόνια. Ως προς τον ε, κύκλο σπουδών και τα μαθήματα καθεαυτά, τον κύκλο μαθημάτων, νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε και να λάβουμε υπόψη το εξή. Εάν μιλάμε για την αυτονομία των πανεπιστημίων που οφείλουμε να τιμήσουμε και εάν θα πρέπει να έχουν και την ευελιξία για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε νέες ανάγκες της αγοράς εργασίας και την παραγωγή νέας γνώσης, είναι δύσκολο να μιλάμε για βασικό κορμό μαθημάτων κάτι το οποίο μας καταδεικνύει και η οδηγία η ίδια. Θα πρέπει λοιπόν τα ίδια τα πανεπιστήμια να δούνε ποια είναι η έκβαση, μάλλον ποιο θα πρέπει να είναι το απότοκο αυτών των σπουδών, αυτού του κύκλου μαθημάτων και αυτό το γνωρίζουν και οι συνάδελφοι μέσω του Tuning Project, το οποίο θα πρέπει να αναπτυχθεί. Υπάρχουν συμφωνίες μερικών πανεπιστημίων σε σχέση με την, ε, το αποτέλεσμα των σπουδών σε κάθε τομέα. Αυτό όμως που δεν έχουμε είναι την, το εφαρμοστικό πλαίσιο στα πανεπιστήμια, το οποίο θα έχουμε σε ένα ε, επόμενο στάδιο. Το πρωί είπατε, κύριε Πρόεδρε, ότι πρόκειται για μια διακυβερνητική διαδικασία και πρόκειται και για μια πρόκληση για την ίδια την έκβαση της διαδικασίας και αυτό με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο, ίσως για διαφορετικούς λόγους. Η συζήτηση βρίσκεται σε επίπεδο κυβερνήσεων εμπολής. Δεν μιλάμε για τα πανεπιστήμια αυτά, δηλαδή, που το μεν μαθαίνει από το δε, θα πρέπει να μεταβούμε σε ένα νέο στάδιο της διαδικασίας της Μπολόνια, όπου θα μιλάμε για επίπεδο εφαρμογής και όχι για εργασία υψηλότερου επίπεδου. Θα πρέπει δηλαδή το πρόγραμμα να εφαρμοστεί με συνέπεια. Ως προς την απασχολησιμότητα των ε, ε, φοιτητών που λαμβάνουν ε, πτυχίο σε επίπεδο δηλαδή και μάστερ και διδακτορικού υπάρχουν προβλήματα ιδιαίτερα σε επίπεδο bachelor διότι υπάρχει διαφορετική μεταχείρισή του. Και πολλά πανεπιστήμια στην ουσία τι κάνουν, ε, επικεντρώνονται, μάλλον συμπυκνώνουν τις ε, σπουδές σε τρία χρόνια, τα οποία αρχικά ήταν τέσσερα. Και γι' αυτό ακριβώς δεν υπάρχει δυνατότητα κινητικότητας αυτών των φοιτητών. Την προηγούμενη εβδομάδα βρέθηκα στο Βερολίνο σε μία διάσκεψη επί του θέματος. Το πρόβλημα αρχίζει να ε, επιλύεται διότι ο κορμός μαθημάτων ε, ξαναεξετάζεται και το HIS στη Γερμανία μετά από μία μελέτη έδειξε ότι πολλοί εργοδότες ήθελαν να απασχολήσουν αποφύτους σε επίπεδο ε, bachelor, κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει στον τομέα της ιατρικής. Υπάρχουν όμως και στους, ε, στον ιατρικό κύκλο σπουδών ε, σημεία εξόδου κατά τη διάρκεια των σπουδών όπου κανείς μπορεί ας να, γίνει, να γίνει υπεύθυνος εργαστηρίου. Έγινε επίσης λόγος για τη συνεργασία με την αντιπέρα όχθη της Μεσογείου. Μιλάμε για συνεργασία και σε αυτό το επίπεδο στα πλαίσια της διαδικασίας της Μπολόνια, με χώρες δηλαδή, με τρίτες χώρες και μετά από τα φετινά γεγονότα, νομίζω ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε τους δεσμούς μας με την ε, αντίθετη όχθη της Μεσογείου. Υπάρχει ένα φόρουμ επαφών μεταξύ των χωρών της Μπολόνια και τρίτων χωρών. Και αυτό προβλέπεται και για τον Απρίλιο του χρόνου στα πλαίσια του Διυπουργικού Συμβουλίου. Θα πρέπει όμως να ενισχύσουμε αυτή τη συνεργασία όχι μόνο σε υπουργικό επίπεδο, αλλά να προωθήσουμε συνεργασία και πέρα από αυτό το επίπεδο, το διυπουργικό, έτσι ώστε νέοι άνθρωποι από την αντιπέρα όχθη της Μεσογείου να μπορούν να έρχονται στην Ευρώπη να σπουδάσουν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και μέσα στα πλαίσια της διαβίου μάθησης προσπαθούμε να καταρρύψουμε το, ε, τα γεωγραφικά εμπόδια ή προσκόμματα στα πλαίσια και της ανώτερης εκπαίδευσης, έτσι ώστε να υπάρχει μια πιο ελεύθερη ροή από τις διάφορες περιφέρειες του κόσμου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Λουίτζι Μπερλιγκουέ και τελευταία παραεμβάση αυτή. Δεν θα είναι η τελευταία, τελευταία ελπίζω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω από βάθους της καρδίας πρώτα απ' όλα την Πρόεδρο για τα λόγια της, ε, για τα λόγια που είπε για μένα. Σας ευχαριστώ ειλικρινά. Ήθελα επίσης να ευχαριστήσω για τη συμβολή όλων των συναδέλφων σε αυτή τη συζήτηση. Όπως είδατε όλοι δείχνουν τεράστιο ενδιαφέρον να συμμετέχουν σε αυτή τη δράση που έχουμε ξεκινήσει και που επιθυμούμε να έχει αποτελέσματα. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι Το τυπικό προβλέπει τροπολογίες και εγώ ειλικρινά επιθυμώ να στις τροπολογίες ε, των συναδέλφων να διαφαίνεται η ίδια δέσμευση όπως αυτή που είδαμε στη συζήτηση. Είμαι πεπισμένος ότι η έκθεση που αυτή τη στιγμή θα πρέπει να έχει μεταφραστεί. Σε λίγες μέρες θα μεταφραστεί και θα είναι έτοιμο. Θα χρειαστεί τροπολογίες, το λέω ειλικρινά. Το γράψαμε ελπίζοντας ότι θα υπάρξουν τροπολογίες και ότι θα υπάρχει μεγάλη συμμετοχή. Ήθελα επίσης να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να ευχαριστήσω τη γραμματεία της ε, Επιτροπής και ειδικότερα την Τερέζα Φαντανέλη ε, αυτής εδώ της Επιτροπής αλλά μιλήσαμε και για την Κομισιόν, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον κύριο Τσάιζεν για την προσωπική του συμμετοχή σε αυτό το έργο. Περνάω στα επιχειρήματα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ξαναδούμε το πρόβλημα της απασχολησιμότητας. Αποτελεί πολύ σημαντικό ζήτημα. Είμαστε όλοι πολιτισμικά πεπισμένοι ότι οι πανεπιστημιακές σπουδέ σίγουρα δεν επιτελούν άμεση επαγγελματική λειτουργία, ωστόσο οι φοιτητέ κάποια στιγμή θα πρέπει να εργαστούν για να ζήσουν και ε, σπουδάζουν για να δουλέψουν. Δεν θα πρέπει όμως έτσι να περιορίσουμε το όραμα που έχουμε για τις σπουδές. Οι σπουδές πριν γεμίσουν ε, το κεφάλι με ένα σωρό ε, θα πρέπει να καθοδηγήσουν τους φοιτητές ε, στο να κατανοήσουν και όχι να γνωρίζουν. Όχι να γνωρίζουν μόνο για να γνωρίζουν, να κατανοούν. Και εδώ έχουμε μία αντιπαράθεση, μία αμφισημία ειδικότερα όσον αφορά τις τρίτες σπουδέ, αλλά και όσον αφορά την τελική φύση του τίτλου υπάρχει και η δυνατότητα να συνεχίσει κανείς θα πρέπει να βρούμε την ισορροπία μεταξύ του, της ε, πολιτισμικής ε, συνιστώσας και της συνιστώσας ε, δυνατότητας εφαρμογής πιστεύω λοιπόν ότι ένα κομμάτι της δυσκολίας ε, Κάποιε δυσκολίε που αντιμετωπίζουν ορισμένα πανεπιστήμια οφείλονται στο γεγονό ότι δεν έχει επιτευχθεί αυτή η ισορροπία. Τα ευρωπαϊκά λοιπόν ειδικότερα κίνητρα και υποδείξει που πρέπει να δοθούν στα κράτη-μέλη και για να αποφασιστεί η αυτονομία και οι ακαδημαϊκοί φορεί που θα πρέπει να διαμορφώσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα πρέπει να βασιστούν σε αυτό, διότι μια διαδικασία όπως αυτή της Μπολόνια η οποία με την απουσία ε, της κυβέρνησης από το σύστημα ε, εάν εγκαταλευθεί μόνο στα, στους ακαδημαϊκούς φορείς ε, εκεί θα επιβληθούν περισσότερο οι επιστημονικές προτεραιότητες. Χρειαζόμαστε λοιπόν να προσφέρουμε αυτό τον εμπλουτισμό στον ευρωπαϊκό χώρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό θα πρέπει να σημαίνει αυτό κατά κύριο λόγο. Κατά μένα είναι πολύ σημαντικό. Εμείς γράψαμε, έχουμε συμπεριλάβει ένα ερώτημα αυτού του είδους μέσα στο κείμενο. Θα σας καλούσα να την ε, μελετήσετε και να την τροποποιήσετε αν χρειαστεί. Το Bachelor είναι το σημείο στο οποίο πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο. αποτελεί καινοτομία εκτός του αγγλοσαξονικού κόσμου και όσοι λένε ότι το Bachelor το τριετές δεν χρησιμεύει σε τίποτα πάνε αντίθετα με την ιστορία. Αυτό δεν είναι αλήθεια σε, καμία, σε κανένα τομέα. Θα ήθελα επίσης να επιστήσω την προσοχή σας στο ζήτημα των ανθρωπιστικών επιστημών, τις φιλολογίες η φιλοσοφία δεν είναι μόνο ανθρωπιστική επιστήμη, ε, είναι και επάγγελμα και επιστημονικό επιστημο, επιστήμη. Δεδομένου αυτού εμείς συμπεριλάβαμε ρητά στο σημείο 11 που θα βρείτε στο κείμενο που θα σας δοθεί στο επίσημο ειδικότερη προσοχή στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων των προγραμματών σπουδών των ανθρωπιστικών επιστημών. Επειδή θεωρήσαμε ότι αυτό θα πρέπει να γίνει σε όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό που ζητάμε εμείς από όσου ασχολούνται με τις ανθρωπιστικές επιστήμες είναι να μας πούν περισσότερο τι αυτό σημαίνει. Ποια είναι η λύση που προτείνεται. Εδώ απλά κατέγραψα το ότι πρέπει να δοθεί προσοχή. Ωστόσο αυτό δεν φτάνει. Γι' αυτό θέλουμε κάποια συμμετοχή, διότι χωρίς ανθρωπιστικές επιστήμες ε, η ανθρωπότητα δεν προχωράει ούτε καν στον κόσμο των επιστημών και της τεχνολογίας. Και εκεί έχει τεράστια σημασία. Επίσης υπάρχει το ζήτημα της γλώσσας. Εγώ είμαι επεπισμένος ε, ότι οι αρχαίοι Έλληνες είχαν καταλάβει τα πάντα από την ανθρώπινη φύση. Ωστόσο η γλώσσα τους δεν έγινε διεθνής ε, γλώσσα. Τα λατινικά έγιναν διεθνής γλώσσα εκείνη την εποχή, στον κόσμο εκείνης της εποχής. Ε, το έλεγε ένας μεγάλος ε, Λατίνος ποιητής. Τα λατινικά έγιναν. Ο Ένιος το είπε. Και στη συνέχεια αυτή τη στιγμή συμβαίνει το ίδιο με τα αγγλικά. Δεν αναγνωρίζω πια τα αγγλικά της, ε, Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι Oxford English. Σήμερα πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτό το διεθνή πτυχή. Πρέπει να το πούμε. Στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια θα πρέπει να υπάρχει κάποιο είδους διγλωσία. Πρέπει να έχουμε το θάρρος να το πούμε. Ακόμη και οι Γάλλοι έφτασαν, κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα σπάζοντας ένα ταμπού. Αυτό μας φέρνει επίσης και στη συζήτηση για τις χώρες εκτός Ευρώπης. Συμμετείχα σε μια συνεδρίαση της ε, ε, Ένωσης Ευρώπης Μεσογείου η Τουνίση, η Τινίση και οι Μαροκινοί μιλούσαν για τη διαδικασία της Μπολόνια στο δικό του σύστημα σε σχέση με το ευρωπαϊκό σύστημα. Υπήρξε ένα πανεπιστήμιο στη Σλοβενία που επίσης συμμετείχε σε αυτό. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτές τις δυνατότητες διεύρυνσης Αυτές είναι περιοχές με ευρωπαϊκή πανεπιστημιακή κουλτούρα. Δεν θα προχωρήσω άλλο γιατί βλέπω ότι η πρόεδρος μου ζητάει να, να ολοκληρώνω. Σας προτείνω λοιπόν να ε, κάνετε τροπολογίες. Αυτό που θέλω να αναφέρω για να ολοκληρώσω είναι το πρόβλημα της αναγνώρισης, το πιο περίπλοκο πρόβλημα, το πιο σύνθετο. Είναι αλήθεια Εντό μιας ίδια χώρας υπάρχουν σήμερα πανεπιστήμια τα οποία δίνουν μάστερ και δεν αναγνωρίζουν τον μπάτσελορ που έχει πάρει κάποιο σε ένα άλλο, άλλο πανεπιστήμιο της ίδια χώρας. Εδώ έχουμε φυσικά πράγματα. Εδώ μιλάμε για την οτροπία του ακαδημαϊκού σώματος που θα πρέπει να καταλάβει την ανάγκη επικοινωνίας επαφής με τους υπόλοιπους. Η αυτονομία είναι ένα καλό πράγμα μεν, αλλά ε, και η συνεργασία είναι καλό. Πρέπει να καταλάβουμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν αντικειμενικοί παράγοντες ε, στα προγράμματα σπουδών. Θα τα μελετήσουμε όλα αυτά όταν θα συζητήσουμε τις τροπολογίες. Ευχαριστώ θέρμα όσους από εσάς ε, είπατε τις απόψεις σας και συμμετείχατε σε αυτή τη συζήτηση. Σας ευχαριστούμε θερμά στα Ιταλικά συνάδελφε Μπερλιγκουέρ, η Πρόεδρος. Στους συναδέλφους θέλω να επισημάνω κάτι. Δεν μπορείτε να συντάξετε τροπολογίε γιατί δεν έχουμε ακόμα έκθεση, εντάξει. Δεν μπορείτε να συντάξετε τροπολογίε. Δεν έχουμε έκθεση στα χέρια μας. Ο κύριος Μπέρλιγκουερ την έκθεση του στις 23 Νοεμβρίου θα την παρουσιάσει. Και αποφάσισα εγώ ότι δεν θα ψηφίσουμε το Δεκέμβριο, αλλά τον Ιανουάριο τελικά θα ψηφίσουμε προς έγκριση. Αυτό επαρκεί πλήρως πριν από τον Απρίλιο, την επόμενη συνάντηση των υπεύθυνων για την Πολόνια Κάτι 23 θα έχουμε λοιπόν την έκθεση. Θα καθορίσουμε στη συνέχεια καταληκτική προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών μέσα Δεκεμβρίου κάποτε και τον Ιανουάριο, 23-24 Ιανουαρίου θα ψηφίσουμε προς έγκριση. Και μπορούμε στις 20 Δεκεμβρίου να έχουμε πάλι, αν θέλουμε, μια σύντομη συζήτηση για όλα αυτά τα θέματα. Εντάξει, σας ευχαριστώ και πάλι πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Είσαστε όλοι εξοικειωμένοι και σε βάθος με αυτά τα θέματα και διαρκώς οι ψηφοφόροι μας μας αναφέρουν αυτά τα θέματα. Κάπως πρέπει αυτά τα προβλήματα να τα αντιμετωπίσουμε με το σωστότερο τρόπο. Περνάμε στο τελευταίο σημείο της σημερινής μας πρωινής μας συνεδρίασης. Παρουσίαση της μελέτης με θέμα καταποκοπήν τέλος ε, περιεχομένου μια ε, παράνομη ανταλλαγή ε, αρχείων κτλ. από τον Αλέν Μεντό. Έχουμε δώσει εντολή για την παρουσίαση. Οι κύριοι βρίσκονται εδώ και πολύ διάστημα εδώ. Α έρθετε μπροστά εσεί οι κύριοι και να μα παρουσιάσετε τι απόψει σα και τα συμπεράσματά σα από αυτή τη μελέτη σύντομα σε ένα τέταρτο. Παρακαλώ. Και μετά στη συνέχεια θα έχουμε άλλο ένα τέταρτο για ερωτήσεις, απαντήσεις και θα έχουμε τη συνάντηση των συντονιστών στη συνέχεια. Monsieur δεν ξέρω ποιος θα ξεκινήσει. Εσείς κύριε Μοντό πρώτος αν λειτουργούν τα τεχνικά θέματα και οι συσκευές ε, και τα λοιπά, ξεκινήσουν. Και αυτό είναι ένα θέμα που είναι και αυτό σημαντικό σίγουρα. Ζούμε σε μια τόσο τεχνολογικά εξειδικευμένη μορφή του σύγχρονου κόσμου με τηλέφωνα, ε, iPod και άλλες συσκευές. Ε, αυτά είναι σημαντικά θέματα. Γι' αυτό χαιρόμαστε που δώσαμε εντολή για αυτή τη μελέτη. Θα μας την παρουσιάσετε αμέσως τώρα εσείς. Ο κύριος Μοντό παρακαλώ, έχετε τον λόγο. In English you are speaking. Yeah. Αγγλικά θα μιλήσετε κύριε, έτσι. Εντάξει, ωραία. Yeah. Merci, merci, Madame la Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσετε στα αγγλικά ή στα γαλλικά. Στα γαλλικά. Ε, ωστόσο η παρουσίαση που έδωσαν ήταν στα αγγλικά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριοι βουλευτές. Ε, με μεγάλη τιμή σας παρουσιάζω αυτή την εργασία μου εδώ. Συνοδεύομαι από δύο μέλη της ομάδας που συμμετείχαν σε αυτή τη μελέτη, τον Ερικ Λαμπέρ, ο οποίο είναι Ιταλός, ενώ δεν ακούγεται από το όνομά του, και η κυρία Φοντανέλ. Αυτή η εργασία Μα ζητήθηκε λοιπόν πριν από πάνω από έξι μήνες από την Επιτροπή Πολιτισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για μια μελέτη σκοπιμότητας για τη δημιουργία ενός καταποκοπήν ε, τέλους ε, περιεχομένου ε, πας δημιουργίας ουσιαστικά ή πας ε, εικόνας αν αφορά τα οπτικοακουστικά μέσα Ποιε ποιες θα ήταν οι συνθήκες για την υλοποίησή του καμε να περιορίσουμε το έργο μας στη μουσική και στα οπτικά-ακουστικά έργα λόγω των τεράστιων διαφορών που υπάρχουν στις αλυσίδες αξίας και στους τρόπους κατανάλωσης σε σχέση με τα υπόλοιπα πολιτισμικά αγαθά όπως τα ηλεκτρονικά βιβλία ή άλλες μορφές ε, δημιουργικών έργων και επίσης ε, κάναμε τη διάκριση μεταξύ της μουσικής και του οπτικοακουστικού διότι έχουν δύο διαφορετικές αλυσίδες αξίας και δύο διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας. Τα κυριότερα θέματα που αφορούν αυτό το content flat rate, το καταποκοπήν τέλος περιεχομένου, αφορούσαν τα κυριότερα τα κυριότερα προβλήματα ουσιαστικά αφορούσαν την διαφορετικότητα των ε, φορέων και των συμμετεχόντων στον τομέα του ψηφιακού, της ψηφιακής οικονομίας τόσο για τα ακουστικά μέσα όσο και για τη μουσική που καθιστούν, θα το δούμε αργότερα, τη συνένεση εξαιρετικά δύσκολη για να μην πω αδύνατη ενώ το διακύβευμα είναι ουσιώδου σημασία ε, για την υλοποίηση του καταποκοπήν τέλους περιεχομένου. Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο έπρεπε επίσης να αντιμετωπίσουμε είναι οι διάφοροι τρόποι διανομής που σήμερα καθιστούν ε, την κυκλοφορία των έργων εξαιρετικά εύκολη και που θέτουν ωστόσο ένα πρόβλημα αν προσδιορισμού του τύπου δικαιωμάτων και συμπεριφορών των καταναλωτών. Αυτή η αλυσίδα αξία λοιπόν έχει ε, ψηφιακή αλυσίδα αξία επιτρέπει τη συμμετοχή νέων φορέων και έχει τροποποιήσει την αλυσίδα αξίας και τη διανομή των αξιών και δυσκολεύει, δυσχεραίνει τη συνένεση. Επίσης ο ψηφιακός τομέας ε, έχει αλλάξει εκβάθρον τον τρόπο κατανάλωσης των πολιτισμικών αγαθών. Θα έλεγα ότι σήμερα, ενώ για πολύ καιρό τα οπτικοακουστικά, οπτικοακουστικός τομέας εξαρτώταν κυρίως από τους παραγωγούς, σήμερα εξαρτάται κυρίως από τους καταναλωτές. Η δημιουργία λοιπόν ενός καταποκοπήν τέλους περιεχομένου επιβάλλει να λάβουμε υπόψη όλα αυτά τα αντικρουόμενα συμφέροντα και θα υπάρξει μια συνένεση ίσως και αδύνατη, δεν ξέρουμε, σε επίπεδο πολιτικό, σε επίπεδο ευρωπαϊκών ε, θεσμικών οργάνων. Μια πολιτική απόφαση συνεπάγεται, όπως εννοείται, να προσδιοριστούν σημεία εύλογα ε, στις αντιρρήσεις των διαφόρων ε, ενδιαφερομένων και αν τελικά καταλήξουμε στο καταποκοπήν τέλος, ε, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα αιτήματα των μεν και των δε. Διαφορετικά θα είναι αδύνατον. Περί τίνος πρόκειται λοιπόν εδώ. Εδώ προσπαθούμε να ε, επιτύχουμε τρεις κοινωνικούς στόχους, τρεις κύριους κοινωνικούς στόχους, τη διασφάλιση μιας σωστής αμοιβή και δημιουργία αξίας για τους δημιουργούς και για ολόκληρη τη δημιουργική κοινότητα το οποίο συνεπάγεται, θα το δούμε είναι εξαιρετικά σημαντικό, συνεπάγεται έναν τρόπο διανομής αυτής της αξίας εξαιρετικά ακριβή και απολύτως διαφανή και σαφή. Θα πρέπει να επιτρέψει τη δημιουργία ενός πλαισίου σταθερού και κατανοητού για τους επιμέρους καταναλωτές και μία από τις συζητήσεις που είχαμε στην ομάδα επικεντρώθηκε στο ότι θα πρέπει να θα πρέπει οι περιστασιακοί ας πούμε φορείς πειρατείας να επανέλθουν σε μια ε, λειτουργία νόμιμη μέσω αυτού του μηχανισμού του flat rate. Για να επανέλθουμε στο ζήτημα της ε, συνένεσης, σε αυτό το πίνακα παρουσιάσαμε τους κυριότερους ε, ενδιαφερόμενους και τα κυριότερα συμφέροντα αυτού του τομέα, ώστε να δείξουμε τι εμείς θεωρήσαμε από τη μελέτη που κάναμε, πρακτικά στον πίνακα αυτό βλέπετε τους πολίτες, τους καταναλωτές, τους δημιουργούς, τις βιομηχανίες περιεχομένου, τις βιομηχανίες τεχνικές και τους φορείς ISP και τις θέσεις τους, σε τι συμφωνούν, σε τι διαφωνούν όσον αφορά τη δημιουργία αυτού του καταποκοπήν τέλους. Θα δείτε ότι οι πολίτες και οι καταναλωτές είναι υπέρ σε μεγάλο βαθμό. Οι καταναλωτές επιβάλλουν το περιορισμό ότι δεν θα πρέπει να είναι πολύ ακριβή αυτή η υπηρεσία. Ε, στους δημιουργούς ε, οι γνώμες διήστανται ε, είναι υπέρ ε, εφόσον ο μηχανισμός τους εξασφαλίζει εισοδήματα με ασφαλή τρόπο αλλά ανησυχούν μήπως εμποδίζει, μήπως εμποδίζει στη δημιουργία των επόμενων έργων η παραγωγή καταλόγων και οι φορείς που διαθέτουν καταλόγους ε, δεν είναι ιδιαίτερα υπέρ. Ε, συζητήσαμε μαζί τους δύο ζητήματα προκύπτουν ότι δεν πρέπει να σκοτώσουμε τους νόμιμες προσφορές που υπάρχουν σήμερα και δεύτερον δεν θα πρέπει να υπάρχουν απαγορευτικά κόστη διαχείρισης. Οι ηλεκτρονικές και τεχνολογικές βιομηχανίες είναι κατά. Και τέλος, οι υπηρεσίες παροχής ίντερνετ, οι ISP, είναι κατά, διότι προτιμούν, διότι ναι μεν δίνεται πλεονέκτημα στις νόμιμες προσφορές, α, αν όμως ε, αυτή η φόρη αντικαταστήσουν άλλους ίσως ε, να θα μπορούσε να υπάρχει περιθώριο για συζήτηση. Όπως βλέπετε λοιπόν το ζήτημα της συνένεσης είναι εξαιρετικά βασικό. Δεν συμφωνούν όλοι οι φορείς. Για να προχωρήσουμε λίγο περισσότερο, κάναμε τη διάκριση μεταξύ του ζητήματος της τιμής, που είναι βασικό ζήτημα, θα καθορίσει την αξία του τομέα, θα καθορίσει επίσης το κατά πώς θα γίνει αποδεκτό από τον καταναλωτή. Εκεί έχουμε τεράστιες διαφορές μεταξύ μουσικής, όπου υπάρχουν ήδη πολλές προσφορές νόμιμες ε, με φόρτωση από το διαδίκτυο. Αναφέρουμε τα Spotify Deezer, αλλά υπάρχουν και άλλα. Αυτό που είναι σημαντικό σε αυτές τις προσφορές, αυτές οι προσφορές θα πρέπει να είναι δωρεάν ή σε ένα πολύ μικρό, με μια πολύ μικρή χρέωση ε, ως μεγαλύτερα ποσά ανάλογα με τον όγκο ε, τηλεφόρτωσης. Εδώ υπάρχουν επίσης διαφορές μεταξύ μουσικής και οπτικοακουστικών ε, μέσων. Για να επανέλθουμε στο ζήτημα επίσης του κατά πόσο θα γίνει αποδεκτό αυτό το τέλος από τον τομέα. Η τιμή δεν θα πρέπει να είναι ούτε υπερβολικά χαμηλή, διότι θα θεωρεί το κατά κάποιο τρόπο ότι τα έργα παρέχονται δωρεάν. Ούτε πολύ υψηλή ωστόσο, ώστε να μπορεί να είναι ανταγωνιστική με τις σημερινές νόμιμες προσφορές. Αυτό το flat rate λοιπόν, αυτή η καταποκοπήν τιμή, θα πρέπει, είναι πολύ σημαντικό να καθοριστεί σωστά, θα πρέπει να αναλυθεί με ακρίβεια. Εμεί κάναμε μια μεγάλη ανάλυση βάσει διαφόρων ε, πληροφοριών που έχουμε για τις διάφορους τρόπους εκμετάλλευσης και βλέπουμε ότι αυτή, αυτό το καταποκοπήν τέλος πρέπει να αποφέρει ότι θα πρέπει να αποφέρει 56-28 εκατομμύρια στη Γαλλία για το οπτικοακουστικό τομέα. Το ζήτημα λοιπόν της ε, τιμής είναι πολύ σημαντική. Είναι πολύ σημαντικό Θα βοηθήσει λοιπόν το P2P και την ανταλλαγή αρχείων ώστε να εξαλειφθεί η πειρατεία. Θα υπάρχει δηλαδή μια ουσιαστικά επέκταση των νόμων προσφορών και το ζήτημα της τιμής ε, υπησέρχεται επίσης όσον αφορά το, η διαχείριση των προσφορών και τη συλλογή των ε, ε, εσόδων. Αυτό το ζήτημα ζήτημα της τιμής ε, θα βοηθήσει να μην ε, υποβαθμιστούν οι σημερινές ε, νόμιμες προσφορές και στο να δοθεί στον καταναλωτή επίσης πρώτα απ' όλα η αίσθηση ότι έχει value for money, αξία για αυτό που πληρώνει, αλλά θα βοηθήσει να δημιουργηθεί και αξία για τον τομέα, διότι ένα σύστημα το οποίο θα κατέστρεφε την αξία του τομέα λόγω της αδυναμίας του ή διότι θα επέτρεπε υπερβολικά πολλές και διάφορες χρήσεις, θα απορρίπτονταν συστηματικά. Γι' αυτό το λόγο η πρότασή μας επιτρέπει μια πρώτη προσέγγιση, ωστόσο είμαστε πολύ προσεκτικοί. Μιλάμε για 4,99 ευρώ με ΦΠΑ στο η γαλλική αγορά. Αυτό θα ήταν ένα παράδειγμα τιμής για αυτό το καταποκοπήν τέλος περιεχομένου για τα οπτικοακουστικά μέσα σε μια τυπική αγορά. Ε, οι προσφορές ας πούμε ε, στη μουσική για παράδειγμα έχουν διαφορετική αξία από τη μία χώρα στην άλλη και διαφορετικές συνέπειες σε, κάθε, σε διαφορετικές συνέπειες σε κάθε χώρα οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Τι τύπο κατά αποκοπή τέλος θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Υπάρχουν διάφορες ε, λύσεις ε, καθώς αναζητάμε τη συνένεση αν προσπαθούμε να εξαλείψουμε τη διαφορά μεταξύ του νόμιμου και του παράνομου και ψάχνοντας να βρούμε κάτι το οποίο θα μπορέσει να προσελκύσει τους καταναλωτές προς, την ε, νόμιμη, προς το νόμιμο σύστημα. Επίσης τονίζουμε ότι αυτό το σύστημα flat rate θα πρέπει να έχει ε, κάποιες δυνατότητες ε, εκτός ενός συστήματος συλλογικής διαχείρισης βασικά θα πρέπει να βασιστεί σε ένα σύστημα συλλογικής διαχείρισης και όλοι οι επίσημοι κατάλογοι θα πρέπει να περιλαμβάνονται στου καταλόγου. Το άλλο σημείο που μου φαίνεται πολύ σημαντικό στη μελέτη σκοπιμότητας και είναι σημαντικό για το Κοινοβούλιο είναι ότι δεν θα πρέπει να χρειάζεται να αρχίσουμε να κάνουμε τροποποιήσεις νόμων και συνθήκων ε, σε διεθνές επίπεδο. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε όσο μπορούμε τα νομικά εργαλεία που υπάρχουν σήμερα. δείξαμε ότι υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο για αυτόν τον τύπο καταποκοπήν που το είχαμε αντιληφθεί από την αρχή, ωστόσο το επαληθεύσαμε και στη συνέχεια. Ας πάρουμε το παράδειγμα της οδηγίας καλωδιακών και δορυφορικών επικοινωνιών. Δεν θέλουμε να δημιουργηθεί μια νέα εξαίρεση, ούτε επιβάλλει υποχρεωτική αδειοδότηση, περιορίζει την άσκηση των αποκλειστικών δικαιωμάτων στην εταιρεία συλλογική διαχείριση. Συνεπώ, τα... αυτή η εταιρεία συλλογική διαχείριση θα έχει τα δικαιώματα η οποία θα αναλάβει την συλλογή των ε, δικαιωμάτων ε, και τα αναδιανέμει σε όσους, στους δικαιούχους. Αυτό το νομικό πλαίσιο λοιπόν είναι συμβατό με τις ε, διεθνείς συνθήκες για το downloading ε, των ε, έργων θα υπάρχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης ανταλλαγής φακέλων υπό συγκεκριμένες συνθήκες και συγκεκριμένους περιορισμούς με τη συμφωνία των δικαιούχων οι οποίοι θα προσφέρουν τα έργα στην ε, μονάδα συλλογικής διαχείρισης. Για να προχωρήσουμε λίγο πιο πολύ στη μελέτη σκοπιμότητας για να ε, περιγράψουμε λίγο αυτό το flat rate, αυτό το καταποκοπήν τέλος. Θα περιορίστε σε ένα τέλος ε, downloading και uploading ε, για αυτά τα έργα τα οποία θα διατίθενται σε ένα δίκτυο ανταλλαγής peer-to-peer, -peer, διωμότιμο, δηλαδή P2P, Επίσης θα πρέπει να περιοριστεί ενδεχομένως ο αριθμός, ε, το πλήθο ανταλλαγών ε, για τους τελικού ε, χρήστες. Έτσι εδώ θα αποκλείονται οποιασδήποτε εμπορικές πλατφόρμες όπου γίνεται επαγγελματική εκμετάλλευση αυτών των ανταλλαγών. Αυτές οι ανταλλαγές λοιπόν θα επιτρέπονται σε περιορισμένο, για περιορισμένο αριθμό ε, ομοτήμων ας πούμε δεν θα μιλήσουμε για οικογενειακό κύκλο εδώ πέρα θα, 50 άτομα είναι πάνω από τον οικογενειακό κύκλο ε, ε, αλλά το, ουσιαστικά είναι κύκλος ας πούμε συναδέλφων ας πούμε ή εταίρων, φίλων όσον αφορά το streaming και τα cyber lockers δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο αυτής της εργασίας επειδή επιβάλλουν άλλα νομικά ζητήματα τα οποία δεν ζητήθηκε να συμπεριλάβουμε στη μελέτη αλλά για τα οποία θα μπορούσαμε ενδεχομένω να συζητήσουμε. Για να επιτύχει ένα έργο σαν αυτό έχουμε προσδιορίσει τα βασικά κριτήρια, την νομική βάση, την ιδιαιτικότητα, την ε, δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής, τη διαχείριση, την τιμή και το μάρκετινγκ. Μιλάμε για 42 παράγοντες επιτυχίας. Δεν μιλάμε για 42 στάδια εδώ, ούτε για 42 συστάσεις. Μιλάμε για ένα σύνολο δεδομένων ε, ε, σημείων τα οποία θα προσέξουμε, τα οποία θα πρέπει να προσέξουμε ώστε να είμαστε σίγουροι ότι θα έρθει εις πέρα σε αυτό το έργο. Όσον αφορά την πολιτική ε, δυνατότητα υλοποίησης, αυτό το σύστημα δεν ακυρώνει, δεν, ε, δεν καταργεί την πειρατεία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αντικαταστήσει ή να υποβαθμίσει τα επιχειρησιακά μοντέλα που υπάρχουν σήμερα. Είναι ένα συμπληρωματικό σύστημα το οποίο δημιουργεί αξία για την κοινότητα των δημιουργών. Η συνένεση, μάλλον τουλάχιστον για να μπορέσουμε να έχουμε όσο το λιγότερο δυνατή αντίθεση σε αυτό, η συλλογική διαχείριση παρέχει ένα πλαίσιο διαχείρισης για το σύστημα και φυσικά ταυτόχρονα είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε να ενισχύουμε την καταπολέμηση της οπτικοακουστικής πειρατείας και όλες τις υπόλοιπες μορφές παράνομων χρήσεων. Πιστεύω ότι αυτά τα δύο συστήματα λοιπόν θα μπορούν να προχωρούν παράλληλα. Η οικονομική δυνατότητα θα πρέπει να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε όχι μόνο το σωστό τέλος, τη σωστή τιμή, αλλά διαφορετικό τέλος για τη μουσική και για τα οπτικά ακουστικά και το σινεμά. Όταν λέμε οπτικά ακουστικά αυτά περιλαμβάνουν και το σινεμά. Θα πρέπει να φροντίσουμε τα κόστη διαχείρισης να είναι συμβατά φυσικά με τις πραγματικές συνθήκες της διαχείρισης, αλλά να είναι και αποδεκτά σε όλη την αλυσίδα αξίας. Γι' αυτό το λόγο πιστεύουμε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό Ωστόσο δεν προλάβαμε, ούτε είχαμε τα μέσα για να το κάνουμε. Θα πρέπει να μελετήσουμε πιο λεπτομερώς ε, αυτή την πτυχή, να υπάρξει μια ε, σε βάθος μελέτη το κόστου διαχείρισης των παρόχων πρόσβασης, των ε, υπηρεσιών συλλογικής διαχείρισης και το ουσιαστικό ερώτημα του παραθύρου εκμετάλλευσης του περιθωρίου εκμετάλλευση. Όπως γνωρίζετε, πολλοί επαγγελματίες και πολλοί δικαιούχοι ε, χρησιμοποιούν και ειδικέ προσφορές με τις ταινίε που βγαίνουν. Συνεπώ κάτι το οποίο θα αντιστοιχούσε μια τέτοια προσφορά θα ήταν απαράδεκτο, αλλά όπως βλέπουμε σήμερα έχουμε ταυτόχρονη έξοδο ας πούμε μια ταινία ε, DVD, ε, αίθουσα κτλ. Θα πρέπει λοιπόν η προσφορά που θα κάνουμε εμείς να λαμβάνει υπόψη και αυτές τις προσφορές και τα ε, χρονοδιαγράμματα. Είναι λοιπόν πολύ σημαντική διαδικασία, δεν μπορούμε να τη χαράξουμε τόσο εύκολα και τόσο γρήγορα. Επίσης το ζήτημα του τρόπου διανομής των εισοδημάτων, επίσης το ζήτημα μιας ενδεχομένου σήμανσης που θα υπάρχουν στις ιστοσελίδες ώστε να επιτρέπονται αυτές οι ανταλλαγές. Επίσης, πολιτική ανάγκη προώθησης του έργου στο μέγιστο αριθμό δικαιούχων, διότι αν το περιεχόμενο δεν υπάρχει, η τιμή θα είναι πολύ ακριβή και η προσφορά δεν θα είναι ελκυστική. Επίσης θα πρέπει να απευθυνθούμε και σε έχουν καταλόγους επίσης ε, ε, να συμμετέχουν στην συλλογική διαχείριση. Πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτό το έργο από τον καταναλωτή έως την ε, δημιουργική κοινότητα είναι σαφές ότι το εργαλείο προώθησης, πώληση, συλλογής δεν μπορεί σε αυτό το επίπεδο να είναι παρά ο, η, υπηρεσία παροχής ε, ίντερνετ, ο ISP που θα μπορούσε να τιμολογήσει μια βάση όπως μια ασφάλεια ζωής όπως όταν αγοράζετε κάποιο ε, προϊόν σε ένα σούπερ μάρκετ πληρώνετε κάποιο φόρο βλέπετε στην ετικέτα ότι υπάρχει η δυνατότητα να καταλάβετε ότι τόσα ευρώ το μήνα θα πάνε σε κάτι δηλαδή εδώ να υπάρχει δυνατότητα να ξέρουμε ότι τόσο κομμάτι είναι το καταποκοπήν τέλος να ξέρει λοιπόν ο καταναλωτής τι καλύπτει το ποσό που θα πληρώνει το μήνα τι είδου ανταλλαγές του επιτρέπονται και να αποφευχθεί να βάζει κανείς online ολόκληρο τον κατάλογο του ίδιου του καταναλωτή. Να μην χρησιμοποιούνται δηλαδή αυτές οι ανταλλαγέ για φυσικές αντιγραφές και για τη διανομή του με φυσικό τρόπο. Ε, θα μπορούσε να υπάρχει ενδεχομένω ένα μηνιαίο τέλο το οποίο θα πληρώνει στον ISP ο καταναλωτή. Αφού συλλεχθούν τα χρήματα πώς θα διοχετεύονται στην αλυσίδα προς τους ε, παραγωγούς, προς τους δημιουργούς. Ε, εμείς πιστεύουμε ότι μία μόνο εταιρεία συλλογικής διαχείρισης θα μπορούσε σήμερα να κάνει αυτού του είδους την εργασία. Θα συλλέγονται λοιπόν τα έσοδα μηνιαία από τους ISP και θα παρέχονται στην εταιρεία ε, συλλογικής διαχείρισης αφού αφαιρεθούν τα ε, οι δαπάνες ε, λειτουργίας ε, του ISP. Οι εταιρείε ISP, υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, απλά χωρίς θα παρέχουν αυτά τα ποσά, θα ελέγχουν το ποιος το τι είδους λήψεις έγιναν. Θα παρέχονται έτσι τα χρήματα στους δικαιούχους των δικαιωμάτων βάσει μιας μεθοδολογίας διανομής που είναι εξαιρετικά σημαντική διότι αυτή αποτελεί το κλειδί για να γίνει αποδεκτό από τους επαγγελματίε αυτό το καταποκοπήν τέλος. Και εδώ επίσης υποδεικνύουμε κάποιες πιθανές οδούς, ωστόσο δεν ε- λέμε τι πρέπει να κάνουμε Ξέρουμε ότι με τα σημερινά παραδείγματα της Αζικοά ε, που υπάρχει στη Γαλλία το ζήτημα της διανομής βρίσκεται πάντα στην καρδιά των συζητήσεων. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί. Θα πρέπει να μελετήσουμε περισσότερο αυτή την πτυχή και να δούμε τι πρόταση μπορούμε να κάνουμε εάν θα μετράμε πάνω στις πωλήσει, εάν υπάρχουν άλλες μέθοδοι που ενδεχομένως ε, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Αυτό είναι ένα σημείο κλειδί το οποίο δεν αναλύσαμε υπερβολικά, ήταν αδύνατο, ωστόσο απαιτεί πολλές συζητήσεις με πολλούς ενδιαφερόμενους. Το μοντέλο για μας λοιπόν είναι η ΑΖΙΚΟΑ, είναι η Ένωση Διεθνούς Διαχείρισης, Συλλογικής Διαχείρισης των Οπτικοακουστικών Έργων. Εδώ πληρώνονται ποσά για την αναμετάδοση τηλεοπτικών σημάτων στα, σε καλωδιακά και δορυφορικά δίκτυα. Εδώ λοιπόν τα χρήματα των συνδρομητών ενός καλωδιακού δικτύου πηγαίνουν προς την Αζικοά και μία-δύο φορές το χρόνο νομίζω η Αζικοά αναδιαμνέμει ε, τα έσοδα βάσει των δηλώσεων των δικαιούχων. Αυτό που μας φαίνεται σημαντικό στο μοντέλο της ΑΖΙΚΟΑ είναι ότι όλοι οι παραγωγοί συμμετέχουν και οι Αμερικάνοι ακόμη. Με τους τεράστιους καταλόγους τους ε, πρόκειται για ένα μοντέλο το οποίο ε, κατά... είχε πολλούς που, την αμφισβή... το αμφισβήτησαν αλλά σήμερα κανένας δεν το αμφισβητεί πλέον όλοι συμμετέχουν και όλοι αποφελούνται από αυτή την, αυτό το δορυφορικό σύστημα. Συνεπώς τα χρήματα που θα αναδιανέμονται στους δικαιούχους θα καλύπτουν επίσης τις αμοιβέ των ερμηνευτών, των δημιουργών. Θα καταβάλλονται λοιπόν σε αυτούς τους ερμηνευτές και σε αυτούς τους δημιουργούς σύμφωνα με τις συμβάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο το ζήτημα που τίθεται είναι κατά πόσο για εμάς στην Ευρώπη επειδή υπάρχει ήδη μια ε, εταιρεία συλλογική διαχείρισης κατά πόσο αποτελεί διασφάλιση για τους δημιουργούς να γίνεται η διαχείριση από μια τέτοια εταιρεία ε, συλλογικής διαχείρισης. Ε, μια έρευνα λοιπόν που μας φαίνεται σημαντική είναι θα πρέπει να δούμε τη διαφορά τιμών μεταξύ μουσικής και οπτικοακουστικών μέσων, τις διαφορές μεταξύ των διαφόρων χωρών φυσικά και επίσης το κατά πόσο θα ήταν αποδεκτό ένα κόστο, ποιο θα ήταν αποδεκτό κόστος λειτουργίας των ε, παρόχων ε, ISP και ποια θα είναι η μεθοδολογία αναδιανομή των χρημάτων. Ε, Ευχαριστούμε. Κύριε Μωρό, ε, δεν έχουμε πλέον παρά 10 λεπτά για συζήτηση. Δίνω το λόγο στην κυρία Τρούπελ ως πρώτη ομιλητή. Ναι, ξεκινώ με τη συζήτηση για τη διαδικασία της Μπολόνια, όπου είχαμε τα θέματα φιλοσοφίας και φιλοσοφικής προσέγγισης. Σε αυτό το θέμα έχουμε ένα φιλοσοφικά και πολιτικά θεμελιώδες ζήτημα. Αφενός βλέπουμε την ψηφιακή επανάσταση που αλλάζει τη ζωή μας. Ο κύριος Μοντό μόλις είπε η ψηφιακή επανάσταση είναι κυρίως χρόνος καταναλωτών και όχι τόσο θέμα παραγωγών. Και αν δούμε εδώ ότι πολλοί καταναλωτές δεν πληρώνουν και έτσι μεσοπρόθεσμα δεν έχουμε δυνατότητα χρηματοδότησης της πολιτισμικής πολυσχηδίας, δεν είναι τότε ένα υφόρο πρότυπο. Όμως πολλά θέματα της προστασίας δεδομένων πρέπει να ληφθούν υπόψη έχουμε την ειδική αντιπαράθεση μεταξύ παλαιών και νέων μονοπωλίων στη ΣΥΠΑ. Hollywood κατά του ε, Google και των προϊόντων που παρέχονται από τέτοιους ε, παρόχους και υπηρεσίες. Τα νέα μονοπόλια όμως εισπράττουν ε, τα έσοδά τους χωρίς να πληρώνουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Ούτε και αυτό όμως είναι αηφόρο πρότυπο. Λοιπόν γενικά, γενικά κατήθεται το ερώτημα. Οι πάροχοι του διαδικτύου πρέπει να ρυθμίζονται λοιπόν διαφορετικά, με διαφορετικό τρόπο από ό,τι σήμερα, ώστε πολιτικά να δεσμεύονται να καλύπτουν τα θέματα δικαιωμάτων. Και έχουμε και τη συζήτηση στον ψηφιακό κόσμο. Τι είναι εμπορικό και τι δεν είναι εμπορικό. Τι είναι εμπορική ή όχι συναλλαγή. Το εμπορικό είναι ε, κάτι που ε, ε, όπως στη Γερμανία πρόσφατα απαγορεύθηκε και στη Σουηδία παλιότερα είχαμε μια συζήτηση μέσω της ψηφιακής επανάστασης. Τι είναι ιδιωτικό, τι είναι δημόσιο. Θα έλεγα λοιπόν πολλά φιλοσοφικά ζητήματα τίθενται εδώ ως θέματα προσέγγισης. Πρέπει να βρούμε απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς που συνέταξαν αυτή τη μελέτη ότι σημαντικά στοιχεία και προβλήματα αποκαλύπτουν που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Σημαντική είναι η προσέγγιση, η θεμελιώδης προσέγγιση ότι πρέπει ένα σύστημα αδειοδότησης ε, να υιοθετηθεί, να εγκριθεί. Δεν ξεκινούν από εξαιρέσεις, λένε άδεια πρέπει να υπάρχει ώστε τους πνευματικούς ιδιοκτήτες, ε, καλλιτέχνες, ερμηνευτές να τους καλύπτει και οι καταναλωτές μέσω συνδρομής να πληρώνουν με βάση τα δικαιώματα μια τέτοια άδεια, ένα τέτοιο πρότυπο. Έτσι θα είναι νόμιμη η συναλλαγή σε ένα συγκεκριμένο κύκλο ε, καταναλωτών που θα αντλούν αυτές τις πληροφορίες, αυτά τα στοιχεία και θα συναλλάσσονται με αυτά. Αυτό χρειαζόμαστε ως κοινωνία. Μια συλλογική διαχείριση. Γιατί διαφορετικά με αδειοδοτήσεις δεν είναι σε θέση κανείς στο νέο ψηφιακό κόσμο αν δεν υπάρχει ένα τέτοιο συνολικό πλαίσιο να ανταποκριθεί κανείς. Υποβάλλονται και συγκεκριμένες προτάσεις. Διαχωρισμός του τομέα για παράδειγμα της μουσικής από τον, τη λογοτεχνία και άλλες προτάσεις. Διερωτώ με, δεδομένη της στα κοινωνικά δίκτυα γίνεται είναι εφικτή μια τέτοια διαχωριστική γραμμή ή θα έπρεπε να υπάρχει ένα πακέτο στοιχείων που θα προσφέρονται και που θα καλύπτονται μια και λογοτεχνία, μουσική δύσκολα διαχωρίζονται. Είναι ένα θεμελιώδες ζήτημα και ερώτημα δικό μου προς εμάς. Αυτή την προσέγγιση την βρίσκετε πιστική εσείς και λειτουργική ή θα έπρεπε ψηφιακά πακέτα να πληρώνουμε και με αυτόν τον τρόπο να έχουμε ας το πω έτσι μια ευφυή διαχείριση να πληρώνονται κάποια δικαιώματα και όποιος έχει ξεπεράσει ένα πακέτο, ε, ένα εύρος πακέτου να πληρώνει κάτι παραπάνω. Δεύτερο, ένας ολόκληρος κύκλος όπου εδώ εμπλέκονται οι ε, άνθρωποι για τις συναλλαγές τους, οι πολίτες για τις συναλλαγές τους στον ψηφιακό κόσμο, ώστε να μπορούν νόμιμα να συναλλάσσονται. Πώς θα καταλήξουμε σε ένα τέτοιο ποσό, δεν είναι αυθαίρετο ίσως, ε? πώς θα μπορούσε να ελέγχεται η συναλλαγή. Θα ήθελα να τα αποσαφηνίσετε αυτά γιατί δεν είναι σαφή και για τους παρόχους στον ψηφιακό κόσμο διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Πώς τεχνικά δηλαδή κάτι τέτοιο θα είναι λειτουργικό. Δεν υπάρχουν προβλήματα προστασία δεδομένων. Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου. Ευχαριστώ. Ναι, καταρχήν θα ήθελα και εγώ και το λέω εσκεμένα και συνειδητά να ευχαριστήσω για αυτή την πρώτη μελέτη για αυτό το θέμα. Συμμερίζω με την άποψη κάποιων εδώ και τη δική σας άποψη ότι πρέπει περισσότερο να εμβαθύνουμε σε αυτά τα θέματα ώστε στους επιμέρους τομείς να τους φωτίσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να καταλήξουμε ενιαία σε συμπεράσματα. Την θεμελιώδη σκέψη πολύ σωστά την παρουσίασε η Helga Trüppel πιο πριν. Για μένα τίθεται το ζήτημα αυτά τα τέλη σε αυτό το πρότυπο που εσείς προτείνατε που θα εισπράσω, θα εισπράσω με ποια κλίδα θα κατανέμονται σε κάποια χώρα ή στου ε, πνευματικούς ιδιοκτήτε και δημιουργού. Υπάρχουν κάποιες ιδέες, κάποιες προσεγγίσεις θεμελιώδεις σε ένα νόμιμο πλαίσιο ανταγωνισμού ή σε ένα ισοδίκαιο πλαίσιο ανταγωνισμού. Το άλλο ερώτημα που τίθεται είναι, εσείς κάνετε λόγο για μια συνύπαρξη. Συνύπαρξη των ε, προσφορών premium, των προσφορών εμπορικών προσφορών και των flat rate προσφορών κατά αποκοπήν. Κατά πόσον αυτά στις προ, ε, επαγγελματικές προσφορές έχουν επίπτωση όσον αφορά την νόμιμη συναλλαγή με τέτοια πνευματικά, ε, το πω έτσι, ε, ε, στοιχεία ιδιοκτησίας. Εδώ έχουμε και την παράνομη χρήση και εκμετάλλευση ε, έργων και προϊόντων και συναλλαγή παράνομη. Πώς μπορούν εδώ να υπάρξουν προτερήματα και ποια προτερήματα υπάρχουν και ποια επιρροή υπάρχει στι υφιστάμενες προσφορές. Έχετε κάποιες μελέτες ή πρέπει να γίνουν μελέτες επιπρόσθετα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Και πάλι ο κύριος Βάτιμο. Και μετά θα πρέπει να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά. Ευχαριστώ και εγώ κρίνω άκρος ενδιαφέρουσα τη μελέτη. Θα ήθελα να υποβάλω μία ερώτηση υποτυπώδη κατά κάποιο τρόπο. Οι συγγραφείς έλαβαν υπόψη το broadcasting, δηλαδή το Sky ε, μεταδίδει εκπομπές συγκεκριμένου περιεχομένου. Ε, αυτοί που ακούν ραδιόφωνο πληρώνουν μία εισφορά και το ίδιο συμβαίνει και με το Sky δεν θα μπορούσατε να βρείτε ένα διαφορετικό πρότυπο. Γιατί δεν μπορείτε να λάβετε υπόψη δηλαδή αυτό το πρότυπο της ε, καταποκοπίνης φοράς ανάλογα με, το, με την μετάδοση. Ο κύριος Μοντό, όπως σας είπα και πριν δεν έχουμε χρόνο, κύριε Μοντό για να απαντήσετε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω και ο συνάδελφος που είναι δίπλο μου, ο Έρικ, θα απαντήσει σε άλλους, σε άλλες ερωτήσεις. Ε, ε, ε, Ως προς τα 50 χρόνια θα πρέπει να λάβουμε υπόψη κατά πόσο αυτό είναι τα 50 είναι κάτι το, ένα δεδομένο το οποίο θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη. Δηλαδή αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε κατά πόσο στα ομότητα τη δίκτυα θα μπορούσαμε να έχουμε 27 ή 28 ομότιμους. Γι' αυτό βάλαμε ένα, το 50 σαν ένα όριο ανάλογα με τις ε, ανταλλαγές που γίνονται στον κόσμο, δηλαδή στις ανταλλαγές ομοτήμων φορέων στο Facebook και αλλού σε άλλα κοινωνικά δίκτυα. Δηλαδή ε, υπάρχουν ε, ε, δίκτυα τα οποία προϋπάρχουν και τα οποία λάβαμε υπόψη. Θα το δούμε, θα δούμε αυτή τη μελέτη. Είναι μια τεκμηρίωση που βρήκαμε σε ένα νέο έγγραφο το οποίο έχει διανεμηθεί. Καθίσταται σαφές ότι σήμερα οι προσφορές premium αποτελούν την ίδια τη φύση του τομέα της, ε, των κινηματογραφικών προσφορών. Ξέρετε ότι έργα αμερικανικά ή μη μπορούν να βγαίνουν στις αίθουσες πρώτης ε, προβολής σε DVD και σε DVD πρόκειται δηλαδή για νόμιμες προσφορές. Και αυτοί που κατέχουν οι κάτοχοι δικαιωμάτων και οι διανομής μπορούν να συνυπάρχουν στο δίκτυο. Υπάρχει μία προσφορά, ας πούμε, τριών ευρώ, όπου ο χρήστης ε, μπορεί να έχει με ε, τρία ευρώ αυτό που θα μπορούσε να λάβει με 5 ή έξι ευρώ. Αυτό όμως αντιτάσσεται στα συμφέροντα του τομέα. Γιατί μιλάμε για πνευματικά δικαιώματα και για επενδύσεις που γίνονται ως προς το περιεχόμενο. Ως προς τους ε, καλλιτέχνες και τους συγγραφείς, ε, θεωρούμε ότι η κλίδα κατανομής βασίζεται στα, στις συμβάσεις που υπάρχουν μεταξύ συγγραφέων, ε, δηλαδή πνευματικών δικαιωμάτων μεταξύ συγγραφέων ή παραγωγών. Και σε αυτή την περίπτωση γίνεται επανακατανομή, δηλαδή διανομή ε, μεταξύ παραγωγών, καλλιτεχνών και συγγραφέων. Είπαμε ότι αυτή η κλίδα κατανομής θα πρέπει να γίνει ευρέως αποδεκτή ε, για τα ποσά που εισπράττονται. Εάν 20 εκατομμύρια Ευρωπαίων ε, πληρώνουν ένα ποσό 4,5 ευρώ, τότε αυτό το flat rate δεν μπορεί να βασίζεται στην κατανομή του ενός τρίτου. Θα πρέπει να υπολογιστεί σωστά και με σαφήνεια για τους παραγωγούς, ε, καλλιτέχνες και συγγραφείς. Δεν ξέρω, Έρικ, κατά πόσο παρέλειψα κάτι. Έρικ, μιλάμε για την δυσκολία του ψηφιακού κόσμου να μετρήσει το περιεχόμενο με βάση τα μεταφερόμενα ε, byte. ο καθηγητής Βάτιμο θα συμφωνεί μαζί μου ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να πούμε ότι ένα ποίημα ενός στίχου ανοίξει, ε, ε, έχει μεγαλύτερη αξία από ένα βιβλίο φιλοσοφικού περιεχομένου 300 σελίδων. Αυτό είναι ένα πραγματικό υπαρκτό πρόβλημα σε σχέση με τα διαβιβαζόμενα, μεταφερόμενα στοιχεία. Ως προς την επανακατανομή έχουμε δύο στοιχεία. Πώς γίνεται μεταξύ των δικαιούχων και ποια κριτήρια ισχύουν. Ένα από τα ουσιώδη στοιχεία είναι τα, τα... η ποσότητα που κατεβάζουμε από το διαδίκτυο. Επειδή μιλάμε για σύνδρομες, τότε ο παραγωγός θα πρέπει να κάνει μεγάλη ε, διαφήμιση έτσι ώστε να κατεβάζονται αυτά τα δεδομένα από τους χρήστες. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Σε σχέση με τη συνδρομητική ε, τηλεόραση ή τηλεόραση με ένα flat rate, αυτός που παρέχει τη σύνδρομη θα πρέπει να διέπεται από μία σύμβαση και θα πρέπει να υπάρχει ένα νόμιμο πλαίσιο μιας κοινωνικής πρακτικής η οποία έχει αναπτυχθεί στο ψηφιακό τομέα. Δεν θα πρέπει όμως να αναστρέψουμε τα οικονομικά δεδομένα στη δημιουργία που διαδραματίζουν το ρόλο του στην παραγωγή. Δηλαδή δεν μπορεί ένα μέσο να καλύπτει τα πάντα. Χρειαζόμαστε μέτρα καταστολής για να μην υπάρχουν καταχρήσεις. Μιλήσαμε δηλαδή. για την συλλογιστική της απελευθέρωσης σε σχέση με την απάτη. Δηλαδή, μιλάμε για το σκοπό του τελικού χρήση και εδώ θα πρέπει να γίνει ένας διαχωρισμός. Ως προς το Sky πιστεύω ότι αυτό το σύστημα επιτρέπει πράγματι διάφορες δυνατότητες, δηλαδή ένα καταποκοπήν ποσό, αλλά μπορεί ο χρήστης να πάρει το ραδιόφωνο, το τηλεοπτικό δίκτυο, δηλαδή όλο το οπτικοακουστικό είναι ένα ε, εκούσιο σύστημα το οποίο μπορεί να γίνει αποδεκτό από την καλλιτεχνική κοινότητα ή τον ε, παραγωγό. Το σύστημα είναι πολύ ιδιαίτερα περίπλοκο και έχω την εντύπωση μαζί με την κυρία Τρούπελ ότι θα πρέπει να το ξανασυζητήσουμε δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο μπορούμε να δούμε διεξοδικά μέσα σε 10 λεπτά. Θα ήταν λοιπόν σκόπιμο να ξαναδούμε την εργασία σας, η οποία ήταν πολύ χρήσιμη. Θα το συζητήσουμε με τους συντονιστές. Πότε θα δούμε το περιεχόμενο αυτό και με περισσότερο κόσμο. Θα μπούμε λοιπόν στις λεπτομέρειες του σχεδίου Τώρα θα συνεδριάσουν οι συντονιστές. Λύε τη συνεδρίαση.